this. Um, thank you very much for coming along. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα στο εργαστήριο για τη δικαιοχρησία. Είμαι η Βίκη Φόρτ και είμαι η πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, Προστασίας Καταναλωτών. Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάστηκα με τον Τένις στην Επιτροπή. Ήταν πραγματικά πολύ δυνατή φωνή Κυρίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από τότε που τον ξέρω, και έχει τεράστια εμπειρία πολλών χρόνων ως μέλος της Επιτροπής. Τον ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Επίση ο Ντένι είναι πρωτοπόρος για πολλούς σκοπούς που κάποιοι έχουν ξεχάσει και συνεχώς υπενθυμίζει στους συναδέλφους των μεγάλων ομάδων του Κοινοβουλίου την ανάγκη που υπάρχει να δούμε το θέμα της δικαιοχρησίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που το κάνατε αυτό σήμερα. Εγώ πήρα αυτή την έκθεση χθε το βράδυ στο σπίτι και ξεκίνησα να τη διαβάζω. Είναι πραγματικά πολύ λεπτομερής μελέτη της δικαιοχρησίας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν ξεκίνησα να το διαβάζω και δεν έφτασα στην σελίδα 130 ακόμα, είναι ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα στις διάφορες χώρες που λειτουργούν πολύ καλύτερα από μοντέλα άλλων χωρών. Και προφανώς υπάρχουν τομείς όπου οι βέλτιστες πρακτικές θα μπορούσαν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό σε διάφορους τομείς να συμβαίνει και βεβαίω αυτό συνδυάζεται και με άλλη, άλλη δουλειά που έχει γίνει. Για τον ε, τομέα του λιανεμπορίου για το σχέδιο δράσης για το λανεμπόριο το οποίο οδήγησε σε σχετική έκθεση του δικού μου προκατόχου για τους ε, νέους τρόπους προώθησης ε, καλύτερων εμπορικών σχέσεων, καλύτερων εμπορικών συμβάσεων σε όσους βρίσκονται στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Είμαι σίγουρη ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα σήμερα το απόγευμα για το πώς ε, εντάσσεται ο τομέας της δικαιοχρησίας σε όλη αυτή την αλυσίδα και γιατί είναι σημαντικός για χώρες όπου οι μικρές επιχειρήσεις δεν φαίνεται ότι δεν νιώθουν να έχουν ε, την ίδια, να έχουν ισότητα όπλων ε, ούτως πίν με μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε παρόντες όλοι σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι τον Τένις που εξασφάλισε ότι θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε αυτό το εργαστήριο και βεβαίως θα πρέπει να βελτιώσουμε, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές ε, για να δούμε ποιοι τομείς λειτουργούν και ποιοι, ποιοι δεν λειτουργούν και βεβαίω να ενισχύσουμε τις ε, μικρές επιχειρήσεις στην ε, εμπορική σκακέρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Βίκη για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι όντω έχουμε κοινέ απόψεις σχετικά με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και κυρίως ό,τι αφορά την καλύτερη νομοθέτηση. Δεν είμαστε υπέρ της απλής συμπολικής νομοθεσίας, δεν είμαστε υπέρ της γραφειοκρατίας και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αυτές είναι που θα μας δώσουν άλλωστε τα πρώτα πρακτικά παραδείγματα. Δεν χρειάζονται επιπλέον κανόνες, αλλά πρέπει να βρεθούν πρακτικές λύσεις. Οπότε, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσους είσαστε σήμερα εδώ φτάνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές Βεβαίω είναι δύσκολο πάντα να έχουμε αρκετούς παρόντες ώστε να ψηφίσουν ε, αυτές τις ε, ημέρες κυρίως, αλλά ε, χαίρομαι που είσαστε σήμερα εδώ. Θα συζητήσουμε αρκετά σήμερα, καταρχάς τον τρέχοντα κανονισμό, για το, τη δικαιοχρασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πολλά πρακτικά παραδείγματα. Έχουμε πολλούς ε, παρισταμένους εδώ που έχουν τη δική τους εμπειρία από το franchising, τη δικαιοχρησία. Και βεβαίως θα δούμε και τη μελέτη που ζητήθηκε από το ε, Τμήμα Πολιτικής Α του Κοινοβουλίου Από πού προέρχονται τώρα όλα αυτά, πώς ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν από την ε, έκθεση που είχαμε γράψει ως απάντηση στο σχέδιο δράσης για το λιανεμπόριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής συζητήσαμε και το θέμα της δικαιοχρησίας. Να είμαι και να είμαι σαφής από την αρχή. Υποστηρίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την γενική μέθοδο δικαιοχρησίας ε, που καθιστά δυνατό, τη, δυνατή την συνεργασία και βεβαίως αποτελεί εμπλουτισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς. Κάτι που λέμε και στο ψήφισμα. Βεβαίως, μας ενδιαφέρει ταυτόχρονα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα πλαίσια της δικαιοχρησίας, των συμβάσεων δικαιοχρησίας και πώς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να συνδυαστεί με τις ε, συμβάσεις δικαιοχρησίας. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την παρουσίαση της μελέτης και μετά θα δούμε ένα ε, Ολλανδικό project από το Υπουργείο ε, Οικονομικών Υποθέσεων από κοινού με τις επιχειρήσεις και ύστερα θα συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες για το ρυθμιστικό πλαίσιο και για το τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν κάποια πρακτικά στοιχεία που πρέπει να σας αναφέρω. Το εργαστήριο αυτό ε, μεταδίδεται ε, στο ίντερνετ. Ε, υπάρχουν και έντυπα, του, αντίγραφα του προγράμματος και οι παρουσιάσεις καθώς επίσης και τα βιογραφικά σημειώματα των ε, προσκεκλημένων μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Βεβαίω θα υπάρξουν ε, τα πρακτικά της συνεδρίασης σε λίγες ε, εβδομάδες και από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορείτε να παρακολουθήσετε από το ίντερνετ το εργαστήριο. Με μεγάλη χαρά λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο στην δόκτωρα Ανέτα Διεβιορόφσκα, Μαγκάλσκα. Δύσκολο το όνομά σας. Είναι από το Πανεπιστήμιο του Όσναμπρουκ. Τώρα είμαι από τη Γερμανία, λέει η εκπρόσωπος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι το μισό μου όνομα. Αλλά δεν θέλω να σας τρελάνω ολόκληρο το όνομά μου. Όπως υπόθηκε ήδη, μας ζητήθηκε από το τμήμα πολιτικής να κάνω μια μελέτη για τη δικαιοχρησία. Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου και πριν σας εξηγήσω τι κάναμε και πώς το κάναμε, θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη εκ μέρους του καθηγητή Σούλτε Νόλκε, ε, ο οποίος κανονικά θα ήταν εδώ, αλλά η γυναίκα του αρρώστησε. Και αντί να πάει στο, στο σταθμό για να πάρει το τρένο, πήγε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν θα είναι παρόν. Θέλω να επιστρέψω στη μελέτη που κάναμε για το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει διάφορα ερωτήματα που αποτέλεσαν τη βάση της ερευνάς μας. Εδώ αναφέρονται οι ερωτήσεις. Καταρχάς, οι επιπτώσεις της ισχύωσης νομοθεσίας στην, στον τρόπο λειτουργίας ή στο καλής ή κακής λειτουργίας της δικαιοχρησίας. Δεύτερον, ο κανονισμό 330 του 210 χρειάζεται κάποιε προσαρμογέ ή χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή από τη μέχρι τώρα. Τρίτον, θα μπορούσαν οι πιθανέ ευρωπαϊκέ λύσει να βρεθούν μέσα από πρωτοβουλίε αυτορυθμιστικέ. Τέταρτον, τα τρέχοντα συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποια είναι που συστήματα που ασχολούνται με τη διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα τη δικαιοχρησία. Ποια είναι αυτά. Και επιπλέον, ποιε επιπρόσθετε δράσει ε, χρειάζονται παραδείγματος χάρη εισαγωγή νέων ενωσιακών εργαλείων. Αυτή ήταν η βάση από την οποία ξεκινήσαμε. Το νομικό τοπίο της έρευνάς μας ήταν διτό. Καταρχάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μόνο τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις μαζικές εξαιρέσεις των 330-200 του 2010. Και το Κοινοβούλιο μας ζητούσε όλος ιδιαίτερος Συζήτηση εκτό μικροφώνου. Okay. <laughs> Thank you. Uh, so the, par the parliament was... Μας uh, ρώτησε τα το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τις μαζικές uh, ή ομαδικές εξαιρέσεις. Αν υπάρχει ε, ανάγκη να κάνουμε κάποιε πιθανέ προσαρμογέ, Ε, τις ρήτρε, ας πούμε, για το μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό, τι επιλογέ αγορά, ε, την πόλη δικαιοχρησία κτλ. Και το δεύτερο επίπεδο ήταν ε, να κοιτάξουμε την εθνική νομοθεσία. Εδώ ασχοληθήκαμε και με τον, ε, το δίκαιο ανταγωνισμού και με το ιδιωτικό δίκαιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μόνο τον κανονισμό που αφορά τη δικαιοχρησία στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Όμως, σε ό,τι αφορά τα εθνικά δίκαια, την εθνική νομοθεσία, ε, ισχύει ε, το ενωσιακό δίκαιο για τον ανταγωνισμό, αλλά τα κράτη-μέλη μπορούν και το κάνουν, να εισάγουν κανόνες ε, στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου. Και φυσικά το δίκαιο του ανταγωνισμού επηρεάζει το ιδιωτικό δίκαιο. Όμως αυτό δεν ανισχύει ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας κάνω μια επισκόπηση του εύρους της έρευνάς μας Κάναμε έρευνα σε νέα νομικά συστήματα του Βελγίου, της Εστονίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ισπανίας. Πώς το κάναμε αυτό, με ερωτηματολόγια. Και τα άτομα αυτά που αναφέρονται στη διαφάνεια μας δώσανε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, δηλαδή. Κοιτάξαμε και το ιδιωτικό δίκαιο και το δίκαιο ανταγωνισμού και την ομολογία, διάφορα δόγματα που υπάρχουν. Οτιδήποτε υπάρχει λοιπόν. Λοιπόν, ε, τα αρχικά δόγματα ή δεδομένα ε, σε τη διαστολή με την ε, πραγματικότητα της αγοράς. Ξέρω ότι μιλάω τώρα σαν ακαδημαϊκός από καθέδρας, αλλά όταν συνειδητοποίησαμε ότι οι αρχικές μας υποθέσεις, ε, μεθοδολογικές ε, υποθέσεις, ήταν λανθασμένες ή μάλλον ήταν διαφορετικές από αυτό που πιστεύαμε αρχικά πριν ξεκινήσουμε ότι θα είναι, χρειάστηκε να προσαρμόσουμε τη μεθοδολογία μας, τον τρόπο εργασίας μας. Και βρήκαμε ότι οι πηγές μας, ή μάλλον είναι δύσκολο να βρούμε υλικό για τη δικαιοχρησία. Φυσικά υπάρχουν ε, πολλοί άριθμες δημοσιεύσεις, αλλά αφορούν κυρίως τι είναι η δικαιοχρησία και πώς θα πρέπει να την ασκήσει, ποια είναι τα ωφέλη, ποια είναι οι κίνδυνη. Όμως αυτές οι δημοσιεύσεις δεν σας λένε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία συναντάει κανείς στην αγορά. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας στην αγορά. Η δικαιοχρησία είναι μια σύμβαση μεταξύ επιχειρήσεων, B2B. Και τα συμβαλώμενα μέρη μέσα σε ένα ε, ήρεμο περιβάλλον ε, νομικών γραφείων, ας πούμε, συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις. Είναι πολύ Δύσκολο να βρει κανείς όμως την πηγή που είναι το, η σύμβαση. Σπάνια βρίσκει καλής, κανείς συμβάσεις οι οποίες συζητάνε το πραγματικό περιεχόμενο της δικαιοχρησίας το οποίο συνάπτεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεκινήσαμε συζητήσεις με τους εκπροσώπους των μερών για να ερευνήσουμε τις πρακτικές. Γιατί δεν είχαμε άλλες πηγές. Εδώ πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις δικαστικές για τη δικαιοχρησία. Και αποφάσεις δικαστικές. Φυσικά τα νούμερα δεν είναι πολύ ψηλά είναι πολύ δύσκολο λοιπόν με βάση μόνο τις αποφάσεις των δικαστηρίων να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή με βάση τα όσα αποφάσισαν τα εθνικά δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που κάναμε, με σκοπό να ετοιμάσουμε αυτή την έκθεση που μας ζητήθηκε, είχαμε πολύ άριθμες συζητήσεις με εκπροσώπους των δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Κάναμε μία-μία έτσι, συνάντηση με δικαιοδόχους, αλλά είχαμε 20 ή 30 συζητήσεις ανεπίσημες και με δικαιοπαρόχους και με δικαιοδόχους. Αντί λοιπόν να κάνουμε ό,τι συνηθίζεται συνήθως για τέτοιου είδους έρευνα, να ελέγξουμε δηλαδή τις πηγές, την τεκμηρίωση, τη βιβλιογραφία, τις υποθέσεις, κάποια επίσημα έγγραφα, εστιάσαμε στις επαφές και στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των μερών, των δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων δηλαδή. Μεθοδολογικός πώς αυτή η έρευνα έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα. Και σε τι καταλήξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας. Ότι σε ό,τι αφορά τη δικαιοχρησία, έχουμε να κάνουμε μια πολύ ειδική σύμβαση ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες συμβάσεις B2B μεταξύ επιχειρήσεων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ε, συμβάσεις ε, διανομής διαφορών τύπων. Έχετε αυτά τα δύο επίπεδα ή στρώματα σχέσεων μεταξύ των μερών που εγκυμονούν πιθανώς προβλήματα. Καταρχάς, η δικαιοπάροχη είναι πιο ισχυρή από τους δικαιοδόχους. Αυτή είναι η κλασική κατάσταση. Μπορεί φυσικά σε μερικές περιπτώσεις ε, να έχουμε κάποιους δικαιοδόχους που είναι πιο ισχυρή από τους δικαιοπαρόχους. Αλλά συνήθως την ισχύ την έχει ο δικαιοπάροχος. Αυτός διαπραγματεύεται ε, από θέση ισχύω, έχει καλύτερες πληροφορίες, καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Όμως, αυτή η διαφορετική ανισορροπία συνδυάζεται και, και με αμοιβαία έκθεση ή ευπάθεια, αν θέλετε, των μερών, έτσι το λέμε. Τι σημαίνει αυτό. Ε, τα μέρη συμπεριφέρονται με μη τυπικό, μη χαρακτηριστικό τρόπο. Δηλαδή, από τη μία, ο δικαιοπάροχος αποκαλύπτει τα εμπορικά μυστικά του. Συνήθως τα εμπορικά μυστικά παραμένουν μυστικά, δεν τα αποκαλύπτει στο άλλο μέρος. Όμως ο δικαιοπάρχο το κάνει ούτω ώστε να πετύχει αυτό που θέλει. Και ο δικαιοδόχος απεμπολεί ένα τμήμα της ανεξαρτησίας του. Και αυτό είναι ε, ατυπική συμπεριφορά για ε, επιχειρηματία, ο οποίος κανονικά πρέπει να είναι εξάρτητος και ελεύθερος να κάνει ό,τι καλύτερο πιστεύει ότι πρέπει να κάνει για την επιχείρησή του. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της δικαιοχρησίας. Και αυτό το πράγμα δεν λαμβάνεται υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον κανονισμό των ομαδικών εξαιρέσεων. Αυτό που συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ότι οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξελίσσονται από ειδικού κανόνες για τη δικαιοχρησία σε... στο να αντιμετωπίσουμε τη δικαιοχρησία σαν ε, οποιαδήποτε άλλη υπόθεση συμβάσεων διανομής. Έχουμε την ε, υπόθεση προνούπτια. Αντιμετωπίστηκε εκεί η δικαιοχρησία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχέσεων μεταξύ των μερών, εκεί, αλλά καθώς ε, προχωρούσε, περνούσε ο χρόνος, ε, ενεργοποιήθηκαν οι μαζικές, ε, ο κανονισμός των μαζικών εξαιρέσεων και εξαφανίστηκε το σημείο αυτό, το στοιχείο αυτό από τα, την παλέτα νομοθετικών μέτρων. Το δίκαιο ανταγωνισμού επηρεάζει τις σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου. Το θέμα είναι πώς. Και αν ναι, πόσο βαθιά τις επηρεάζει και ποιες είναι οι συνέπειες. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν λαμβάνεται αυτό το στοιχείο υπόψη αρκετά. Έχετε τον κανονισμό μαζικών εξαιρέσεων που έχει μια πολύ ειδική σχέση για, τις, για το, τις σχέσεις, ειδική σημασία για τις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Τα κράτη-μέλη άρχισαν να τη δρούν όμως σε τέτοιου τύπου λύσεις. Γιατί γενικώ πώς το δίκαιο του αγωνισμού αφορά τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς, της καλύτερης ανάπτυξης αγοράς. Ανάμεσα στα δύο μέρη εδώ στη δικαιοχρησία έχουμε τον δικαιοπάραχο που είναι ο πιο ισχυρός. Αυτός είναι που θέτει τους όρους. Αυτό όμως που συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την Πολωνία, τα κράτη-μέλη είναι ότι αρχίζουν τα κράτη-μέλη να αντιδρούν στην αγορά δικαιοχρησίας και προσπαθούν είτε να εισάγουν ήπια μέσα δικαιο, ε, ή να αναπτύξουν νομολογία για να υποστηρίξουν και να επιλύσουν υποθέσεις δικαιοχρησίας. Υπάρχει μια ληστωτή αντίδραση, αυτό συντοπίσαμε. Το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού προσπαθεί να άρει τους φραγμούς ούτως ώστε να αναπτυχθεί καλύτερα η αγορά. Όμως, το παράδοξο είναι ότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχει υποστήριξη προς τον πιο αδύναμο μέσω νομοθετικών λύσεων που δημιουργούν όμως φράγματα και εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Το συμπέρασμά μας λοιπόν ήταν είναι ότι οι αγορές καταρχάς είναι πολύ διαφορετικές, πολύ διαφοροποιημένες μεταξύ τους και αυτό δεν αφορά μόνο τα παλιά κρατημέλη σε αντιδιαστολή με τα καινούρια κρατημέλη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν, υπάρχει μια 20 ετία που χωρίζει τα παλιά από τα νέα κρατημέλη. Τα νέα κρατημέλη αρχίσαν πολύ πιο πρόσφατα να αναπτύσσουν. Και από τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις που είχαμε με τους ε, ενδιαφερομένους, συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο, διαφορε... δύο είδη σχέσεων δικαιοχρησίας στην αγορά και οι διαφορές μεταξύ των σχέσεων αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, ε, στην εκπροσώπηση των μερών υπάρχει έλλειψη ισορροπίας. Οι δικαιοπάροχοι εκπροσωπούνται καλύτερα από τους δικαιοδόχους. Το καταλαβαίνουμε το γιατί βέβαια. Οι δικαιοπάροχοι έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πόρους, ενώ οι δικαιοδόχοι έχουν μικρότερη πρόσβαση, είναι συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ασχολούνται με την, με την καθημερινότητα της επιχείρησής τους. Τρίτο συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε πιστικά επιχειρήματα που υποστηρίζουν τις σημερινές επιλογές του δικαίου ανταγωνισμού. Δεν υπάρχουν. Ε, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοια επιχειρήματα, δεν παρουσιάζονται. Και το τελευταίο συμπέρασμα ήταν ότι είναι σαφές ότι το περιεχόμενο των των περιορισμών, όπως επιτρέπει ο κανονισμός ομαδικών εξαιρέσεων, θέτει κάποια πρότυπα για το ιδιωτικό δίκαιο. Αν κάτι, λοιπόν, μια συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπεται από τον ε, κανονισμό ε, ομαδικών εξαιρέσεων, θεωρείται ως πρότυπο και μπορεί να γίνει δεκτό. Και δεν επαληθεύεται καθόλου σε εθνικό επίπεδο μέσω της εφαρμογής του ε, στις συμβάσεις δηλαδή για άδικους ή παράνομους όρους ή καταχρηστικούς όρους. Οι συστάσεις μας ήταν λοιπόν ότι πρέπει να ενισχύσουμε την αυτοεκπροσώπηση των δικαιοδόχων, λαμβάνοντας υπόψη την εστίαση που μας ε, έθεσε το Κοινοβούλιο, για το θέμα της αυτορύθμισης. Αν υπάρχει αυτορύθμιση, ε, θα πρέπει τα μέρη να εκπροσωπούνται ισότιμα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγχονται οι τα δεδομένα, οι συνθήκε αγοράς. Αυτή η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε για την έρευνά μας δεν μας επέτρεψε να το κάνουμε όμως αυτό και προτείνουμε α, ανώνυμα σημεία επαφής, με τα οποία θα έρθουμε σε επαφή δηλαδή, ε, για να διερευνήσουμε τι γίνεται στην αγορά. Για να δούμε σε ποιο βαθμό όλε οι εικασίε που έχουμε γύρω από το δίκαιο ανταγωνισμού είναι σωστέ και ποιε είναι οι επιπτώσει του ε, στις στι σχέσει ιδιωτικού δικαίου. Και με βάση τις πληροφορίες που θα έχουμε συλλέξει, περαιτέρω δράσεις μπορεί ε, να είναι καλό να αναλυθούν. Ξεπέρασα και το χρόνο μου κατά δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, ε, Aneta. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ανέτε. Ανέτα. Και ξέρω ότι είναι πολλέ οι μελέτε που κονούνται στο Κοινοβούλιο, όμω η δική σα έκθεση ήταν ιδιαίτερη. Έπρεπε να ασχοληθείτε και να μιλήσετε απευθεία με του ενδιαφερομένου εσεί και να βασιστείτε σε μεγάλο βαθμό στην πείρα και τις ζυμώσεις που προέκυψαν από τις συζητήσεις σας με τους ενδιαφερομένους. Νομίζω ότι είπατε κι εσείς, χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες εξηγήσει για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εδώ θα πρέπει να δούμε τη συνέχεια της συζήτησης και να δούμε τις πολιτικές επιλογές ιδίως για το μέλλον. Μέρος του ε, διαλύματος για τις διακοπές θα το περάσουμε συντάσσοντας μια έκθεση πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβουλίο για το θέμα αυτό που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνη και για την, ανταγωνιστική, για την πολιτική ανταγωνισμού. Και όπως είπατε, ε, πολλά θέματα της πολιτικής ανταγωνισμού έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να δούμε τι τράση θα αποφασίσει να αναλάβει σχετικά το Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη μου χαρά που εν τέλει είχαμε κάποιον Υπουργείο Οικονομικών, α, υπεύθυνη για τα θέματα οικονομικών, την κυρία Φράντσιν, διότι το Ολλανδικό Υπουργείο ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον κώδικα δικαιο, ε, δικαιοχρησίας στην Ολλανδία και μελέτησε πολύ προσεκτικά τον όλο τομέα. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιόγκα. Στι κάτω χώρε ασχολούμαστε με το θέμα τη δικαιοκρασία εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε ε, το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων άρχισε να ασχολείται με την προσέγγιση μα σχετικά, αλλά άρχισε να δίνεται και μεγάλη προσοχή από τα μέσα μαζική ενημέρωση και τα δικαστήρια, διότι υπήρχαν εντάσει μεταξύ δικαιοπαράγων και δικαιοχρηστών. Ε, εδώ. Ε, ασχοληθήκαμε ε, με το νομικό σκέλος του θέματος, αποφασίσαμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέσα σε λίγους μόλις μήνες, το 2015, είχαμε συνεντεύξεις με δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους, ε, με παρόχους νομικών υπηρεσιών και τους ε, πελάτες τους, για να δούμε πού είναι τα προβλήματα και πού προκύπτουν οι δυσκολίες. Είχαμε αρκετέ διαγνώσει. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο βαθμό απάτη, δηλαδή η δικαιοχρησία χρησιμοποιείται ω βιτρίνα και κάποιοι ε, καταχρώνται του συστήματο των δικαιοχρησιών. Κάποιε φορέ είναι επιχειρηματίε, άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά του, έχει πτωχεύσει η επιχείρησή του και χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα προσπαθώντας ε, με εξαπάτηση να εκμεταλλευτούν το όλο σύστημα. Έπειτα στον πραγματικό κόσμο των δικαιοχρησιών με τις πραγματικές ε, και τα γνωστά χαρακτηριστικά του όλου θέματος ε, καθορίζονται διαφορετικές φιλοδοξίες και στόχοι μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε διαφορετική ε, ε, κατανομή των εξουσιών μεταξύ δικαιοχρηστών ε, και δικαιοπαρόχων. Οι περιπτώσεις απάτης έχουν να κάνουν με το ότι ο δικαιοδόχος έχει πολύ διαφορετικές προσδοκίες και σχέδια όταν περνάει στη σύμβαση και τελικά αυτά δεν εκπληρώνονται. Βλέπουμε να υπάρχει μεγάλος βαθμός καχυποψίας και μεταξύ των δύο πλευρών και στο όλο σύστημα κυρίως μεταξύ των ε, νομικών, των παρόχων νομικών υπηρεσιών και των ε, πραγματικών υπηρεσιών. Υπάρχουν ε, δυσκολίε βέβαια ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα και εξαιτία αυτών των δυσκολιών αποφασίσαμε να οργανώσουμε συζητήσει τρογγυλή τράπεζα και να δούμε τι επιλογέ υπάρχουν για την σειρά με την οποία εξετάσουμε τα διάφορα προβλήματα και να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε και να ε, τα καθορίσουμε. Εδώ αποφασίσαμε ότι η απάτη είναι ένα πρόβλημα για όλους, είναι ένα θέμα της βάσης της συνεργασίας μας και προκειμένου να ε, δώσει την απαραίτητη σημασία ο εισαγγελέα, ε, πρέπει να επισημάνουμε και εμείς τα ανάλογα θέματα. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί πρώτο γιατί διαρκώ ανακύπτει στι συζητήσει για τα πραγματικά προβλήματα δικαιοχρησία. Αυτό έπρεπε λοιπόν να βγει από τη μέση. Το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο γύρο συνεντεύξεων ήταν ε, πολύ ευρύτερο, με 60 άτομα τουλάχιστον, δικαιοδόχους, δικαιοπαρόχους, ε, παρόχου, νομικών υπηρεσιών και το Είχαμε αντελεχεί συζητήσει για να δούμε πού πρέπει να φτάσουμε στο όλο σύστημα το 2020. Το συμπέρασμα ήταν ομόφωνο. Ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για την αυτορύθμιση, πρέπει να καταρτηθεί ένας εθνικός κώδικας και πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος κώδικας ανατομέα. Επίσης, ότι χρειάζεται και ένα εξοδικαστικό σύστημα επίλυσης διαφορών, διότι οι δικαστικές ε, διαδικασίες δεν είναι αρκετά σκόπιμες για να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις στο όλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων, βάσει αυτών των αποφάσισε να προβλέψει ένα κονδύλι από τον προπολογισμό, δύο υπαλλήλου ε, για να αναλάβουν να συντάξουν το σχετικό κώδικα. Ε, κάναμε μια προκήρυξη για υποψηφιότητε για τη σύνταξη του κώδικα και η Ένωση για τι Δικαιοχρησίε μα πρότεινε εκ μέρου των ε, δικαιοπαρόχων δύο υποψηφίου, ίδια και από την πλευρά των δικαιοδόχων, για να υπάρξει πλήρη εκπροσώπηση στην Συντακτική Επιτροπή. Τα μέλη αυτά ήταν εθελοντές, δεν υποχρεώθηκαν, ε, ήταν στον ελεύθερο χρόνο τους γιατί αμυστή ε, προσέφεραν τι υπηρεσίες τους, οπότε έκαναν πάρα πολύ δουλειά. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε και τους διάφορους ε, συμβούλους από think tank που μπορούσε να, στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση. Και το πρώτο σχέδιο της έκθεσης καταθέθηκε σε πλήρη εμπιστευτικότητα για να αποφασίσουμε να είναι ένα συνεκτικό, γιατί αποφασίσαμε να είναι ένα συνεκτικό σύνολο πρωτόκολλο στο Έξι μήνες χρειάστηκε να συνταχθεί ο κώδικας δικαιοσύνης για την Ολλανδία και λάβαμε 150 σχόλια για τον κώδικα αυτό εκ των υστέρων, τεράστιος όγκος για τέτοιου είδους κώδικα και από την πλευρά των δικαιοπαράχων και των δικαιοδόχων. Η αντίδραση των δικαιοδόχων ήταν ε, εντάξει, καλά, να συνεχίσετε ενώ ήταν πιο τεχνική η τοποθέτηση των δικαιοπαρόχων, ε, με περισσότερο λεπτομερείς νομικές παρατηρήσεις. Όλα αυτά πραγματικά μας διευκόλυναν για να βελτιώσουμε τον κώδικα αυτόν καθ' διότι η πρώτη εκδοχή ήταν απλώς ένα πρώτο, ε, μια πρώτη εκδοχή των πορισμάτων μας. Ξαναπήγαμε λοιπόν στη Συντακτική Επιτροπή για να τον βελτιώσουμε, ξαναγράφοντάς τον και διορθώνοντας. Έπειτα, είδαμε να υπάρχει και βία απόρριψη από ένα μέρος ε, των ε, δίκαιο παρόχων. Αρκετά βίαιες αντιδράσεις. Προέκυψαν λοιπόν κάποια ζητήματα τα οποία τα ξανασυζητήσαμε για να δούμε αν πραγματικά είναι προβλήματα και σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε ότι είναι όντως προβλήματα, προσαρμόσαμε ανάλογα τον κώδικα, αλλά πιστεύω ότι καταλήξαμε σε ένα πολύ εξισορροπημένο σύνολο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει φόβος περιορισμών των ελευθεριών να ε, αναπτύξει κανείς τις δραστηριότητε που θέλει, να αποκομίσει κέρδος, αλλά ο στόχος δεν ήταν να επηρεάσουμε τη διαδικασία, ήταν σε ένα κλάδο που και δύο πλευρές χρειάζεται να συνεργάζονται και είναι καταδικασμένες οι δύο πλευρές να συνεργάζονται, να γίνεται αυτό με τρόπο δίκαιο, με όρους ισότιμους. Πολλοί ήταν και οι οι οποίοι κοίταξαν πολύ προσεκτικά τι συμβάσει δικαιοχρησία του για να δουν αν ε, συνάδουν με τον κώδικα και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Αυτό μα έδωσε αρκετέ ε, ελπίδε για το μέλλον. Ότι όταν οι δικαιοπάροχοι αρχίσουν να εξετάζουν προσεκτικά τον κώδικα θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Και αυτό δεν μα εξέπληξε, διότι τον κώδικα τον ε, συνέταξαν και δικαιοπάροχοι και δικαιοδόχοι ταυτόχρονα με τι ανάγκε και των δύο υπόψη. Ο κώδικα λοιπόν αυτό είναι ένα όργανο αυτορύθμιση, πολύ ευέλικτο, με κάποιε γενικέ κατευθυντήρε γραμμέ για το πώ να διοργανωθούν οι δικαιοχρησίε, αλλά προσαρμόζεται στου διάφορου κλάδου, τα είδη ενώσεων, το μέγεθο των ομίλων που παίρνουν μέρο ή μπορεί να καλύπτονται. Κάποια πράγματα που συμπεριλαμβάνει ο κώδικα είναι απαιτήσει διαφάνεια, που είναι πολύ σημαντικέ στην φάση τη ε, σύναψη τη σύμβαση τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει μια σύμβαση και γενικού προσανατολισμού για το πώ αυτά να καταρτίζονται. Επίση, ασχολείται με τι διαδικασίε για την συλλογική λήψη αποφάσεων και ε, περιέχει κατευθυντήρε γραμμέ για την ε, πάυση, τη λήξη τη ε, σύμβαση δικαιογραφία με σεβασμό των συμφερόντων και των δύο πλευρών. Ο κώδικα βασίζεται σε αρχέ ε, λήψης αποφάσεων με βάση την λογικότερη επιλογή με συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συλλογική λήψη αποφάσεων βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας και με συνολικές απαιτήσεις ε, διαφάνειας που είναι πολύ σημαντικές. Για την εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών είδαμε τις επιλογές που υπήρχαν μαζί με τη Συντακτική Επιτροπή και ε, δείξαμε ένα πρωτομοντέλο μοντέλο αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ίδιο ο κλάδο θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου που να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ω ε, πηγή για να δουν τι ανελακτική επίλυση διαφορών θέλουν. Οι αριθμοί αυξάνονται ε, και θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνεννοηθούν για να σχηματίσουν αυτή την πλατφόρμα. Ωστόσο και το Υπουργείο μας είχε, είχε καταστήσει τελείως σαφές ότι ε, εάν στην νομοθεσία δεν επιτελεστεί παρκή πρόοδο, η αυτορύθμιση θα πρέπει να προέχει. Τους ερχόμενου μήνε θα δούμε τι θα απογίνει. Σα ευχαριστώ πολύ. Νομίζω η αγγλική εκδοχή του Ολλανδικού κώδικα δικαιοχρησίας είναι διαθέσιμη στην αίθουσα. Εάν το δείτε, είναι μια πολύ μετάβαση από την μια παρουσίαση στην άλλη. Διότι ο κώδικα αυτός τη δικαιοχρησίας αναφέρεται στις ανάγκες του εμπορικού δικαίου και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα πρώτα στάδια σύναψη σύμβαση. Βλέπουμε λοιπόν τι συσχετισμό υπάρχει από τη μια από τις ανάγκες της πρακτικής και την άλλη Τη θεωρητική τοποθέτηση των ε, υπευθύνων των μελετών. Τώρα έχουμε το δεύτερο πάνελ με τον κύριο Χέντριξ, τον κύριο Τσόπρα και τον δόκτορα Άμπελ. Παρακαλώ ας έρθουν για το πρώτο πάνελ.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 παρέμβαση, αλλά θα έρθω μετά σε αυτή. Ε, ο πρώτος ομιλητή στον καταλογό μου είναι ο κύριο Λουκ Χέντριξ, τον οποίο ξέρουμε πολύ καλά, από την ε, UEAPME, την, ε, τον οργανισμό, τον, την οργάνωση ομπρέλα των Ευρωπαίων Εργοδοτών και θα του δώσω κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ. Ντένις, καταρχάς Ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Η δικαιοχρησία, από ό,τι φαίνεται, γίνεται πολύ δημοφιλές ε, θέμα ε, μετά από 20 χρόνια σιωπής. Ξαφνικά κάποιοι εντόπισαν ότι υπάρχουν προβλήματα και είμαι ευγνώμων στον Ντένις που οργάνωσε σήμερα αυτό το εργαστήριο. Ήδη αναφέρθηκε ότι εγώ ε, εκπροσωπώ την UEAPME. Ε, Γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν είμαστε μια οργάνωση που απλώς παραπονιέται ή που απλώς ε, προσωπεί μια μικρή ομάδα δικαιοδόχων. Όχι, είμαστε η οργάνωση που προσωπεί τους εργοδότες μικρομεσαίων των, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκπροσωπούμε λοιπόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στο λιανεμπόριο, αλλά σε όλα τα είδη, σε όλους τους τομείς εμπορίου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Κυρίως εσείς όταν ακούσετε τα σχόλιά μας. Και επίσης, εκπροσωπούμε 12, 12 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλο ένα που ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι ως ε, ε, ως οργάνωση είμαστε θετικά διακείμενοι απέναντι στην ε, ε, δικαιοχρησία κυρίως γιατί τώρα για να είναι κανείς στη σημερινή εποχή ανταγωνιστικός ως μικρομεσαία επιχείρηση ή ως εργοδότης πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο. Κυρίως στον τομέα της, του λιανεμπορίου όπου υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός, παγκοσμιοποίηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντα έχουν περιορισμένους πόρους οπότε ένας από τους ε, ε, τρόπους να λύσουμε το πρόβλημα αυτό είναι να συνεργαστούμε μέσω ας πούμε της δικαιοχρησίας. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Η καλή εμπορική συνεργασία εξαρτάται από τις προσπάθειες και των δύο μερών. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Και τα δύο μέρη πρέπει να κάνουν την απαραίτητη προσπάθεια. Βεβαίω υπάρχουν διάφορες φόρμουλες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η δικαιοχρησία φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ήδη από την δεκαετία του 80 στην, για το λιανεμπόριο, υπήρχε βεβαίω από πιο πριν, αλλά από τη δεκαετία του 80 και από, την, από το πρώτο νομικό πλαίσιο που υπήρξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 88, υπήρξε μία τάση ή δικαιοπάροχη να ε, επιβάλλουν μονομερείς διατάξεις στις ε, συμβάσεις δικαιοχρησίας τους. Εκεί πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μιλούμε για έναν ε, δικαιοπάροχο και έναν ελεύθερο επαγγελματία. Ο δικαιοδόχος παραμένει υπεύθυνος για την εκμετάλλευση. Οπότε είναι σημαντικό να έχει το χώρο για να εμπλακεί προσωπικά και να αναπτύξει τις ιδέες του και τον ε, τρόπο πώλησης του προϊόντος. Και επίσης, ε, πολλές φορές ένα πρόβλημα στις συμβάσεις αυτές είναι ότι δεν υπάρχει χώρος για να προσαρμοστεί το ε, σημείο που θα, η μέθοδος πώλησης στην τοπική αγορά. Και βεβαίως οι συμβάσεις αυτές πρέπει να σέβονται και την ανεξαρτησία και των δύο μερών. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι κάποιες συμβάσεις ήταν ε, ψευτοσυμβάσεις ε, ίδιας απασχόλησης. Αυτό που κυρίως ε, βλέπουμε είναι παλιά προβλήματα που παραμένουν. Δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά, είναι προβλήματα 30 ετών. Αλλά δυστυχώς ποτέ δεν ακούστηκαν τα παράπονα των δικαιοδόχων και των ε, οργανώσεών μας. Στις περισσότερες από αυτές τις συμβάσεις υπάρχει μια υποχρέωση μη ε, δημοσίευσης. Και μάλιστα πάει τόσο μακριά που ο δικαιοδόχος δεν μπορεί καν να ζητήσει συμβουλή από την οργάνωσή του ή από κάποιο νομικό για το περιεχόμενο της σύμβασης πείτε μου ποιος είναι τόσο τρελός που να υπογράψει μια σύμβαση που θα τον δεσμεύει για κάποια χρόνια χωρίς να πάρει την νομική συμβουλή του, των ειδικών. Αυτό λοιπόν υπάρχει. Μετά υπάρχει αυτός ο παράγοντας του κινδύνου, αναφέρθηκε στην έκθεση. Γιατί από τη στιγμή που ε, υψώνει κάποιο τη φωνή του, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Και μετά αρχίζει, ε, αρχίζει η άλλη μεριά να ποινικοποιεί, να λέει ότι εσείς δεν σέβεστε τη σύμβαση, εσείς δεν είστε καλός επιχειρηματίας, εσείς δεν κάνετε αρκετά. Αυτό ε, ισχύει και παλιά, συνεχίζεται, συνεχίζει να ισχύει και τώρα. Τη στιγμή, αυτή τη στιγμή ξεκινήσει κάποιος να αντιδρά. Γι' αυτό πολλοί ε, είναι αρκετά κινούνται αρκετά συντηρητικά στο να πάνε στις οργανώσεις τους. Και επίσης υπάρχει και ελάχιστη νομολογία και υπάρχει και ελάχιστη βιβλιογραφία σχετική. Καταρχάς, λόγω αυτού του παράγοντα, λόγω αυτού του φόβου, γιατί αν πάει κανείς στο δικαστήριο, ε, ξεχάστε το, ούτως ή άλλως κοστίζει και πάρα πολύ. Και μετά το θέμα είναι ότι η νομική βιβλιογραφία τις περισσότερες φορές έχει γραφτεί από νομικούς που είναι οι νομικοί των δικαιοπαρόχων. Οπότε η νομική βιβλιογραφία που υπάρχει, η, ε, στη νομική ε, βιβλιογραφία που υπάρχει, την χάνουν υπεράσπιση στα δικαιώματα των ε, δικαιοπαρόχων. Επίσης, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις για τους δικαιοδόχους σε σχέση με τους δικαιοπαρόχους. Και επίσης, υπάρχει ένα σαφέ συμπέρασμα, ήδη που προέκυψε από την δεκαετία του 90, η προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα, να κάτσει κανείς γύρω από ένα τραπέζι μαζί με τους δικαιοπαρόχους, μαζί με τους δικαιοσδόχους, να συζητήσουν τα θέματα μέσω αυτορύθμισης, απέτυχαν. Απέτυχαν οι προσπάθειες αυτές το δεκαετία του 90, απέτυχαν το 2000 και μετά και θα συνεχίσουν να αποτυγχάνουν. Σε κάποιες χώρες υπάρχει η σχετική νομοθεσία, ας πούμε στο Βέλγιο υπάρχει μια υποχρέωση προσυμβατικής ενημέρωσης Οι επιχειρηματίες λοιπόν που δεν έχουν ενημερωθεί για τις συνέπειες του, της σύμβασης μπορούν να μην την υπογράψουν. Επίσης, δεν δίνεται σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τέτοια θέματα παρό, παρά τις προσπάθειες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς. Ίσως να είναι δικό μας, δικό μας φταίξιμο. Δεν πιέσαμε αρκετά. Τώρα, το θέμα της μη δημοσίευσης, η ρήτρα, η του μη ανταγωνισμού, για την ρήτρα αυτή συνήθως βασίζεται στο ότι υπήρξε μεταφορά τεχνογνωσίας. Το πρόβλημα είναι ότι το περισσότερο καιρό δεν υπάρχει μεταφορά ή υπάρχει ελάχιστη μεταφορά τεχνογνωσίας. Και αν υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας, ο δικαιοδόχος την έχει πληρώσει. Γιατί πληρώνει τέλος. Και σε κάθε περίπτωση, κυρίως στο λιανεμπόριο, στα τρόφιμα ας πούμε, οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτοαπασχολούμενοι ή είναι καινούργοι ή έχουν ένα μικρό μπακάλικο. Ήδη λοιπόν είχαν την τεχνογνωσία. Γι' αυτό πάνε στον δικαιοπάροχο. Τότε πάνε στον δικαιοπάροχο. Δεν νομίζω ότι ο δικαιοπάροχος μπορεί να έχει τόσο μεγάλη πια μεταφορά ή υπερβολική μεταφορά τεχνογνωσίας προς ανθρώπους που ήδη έχουν εμπειρία στον τομέα. Επίσης, στη σύμβαση η αξία της επιχείρησης καταδεικνύεται στην αρχή της σύναψης της σύμβασης, σε περίπτωση που χρειαστεί να απολυθεί στο τέλος. Δεν είναι ισόρροπο λοιπόν αυτό η προσθέμενη αξία που δημιουργείται στην, στην επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργία τη ε, μπορείτε να την ξεχάσετε. Επίση, για τι υπόλοιπε υποχρεώσει. Είναι, πολύ ε, ε, εξαιρετικά περιορισμένη η εμπορική ελευθερία. Επίση, υψηλέ τιμέ που πρέπει να πληρώσει ο δικαιοδόχο. Έχω δει συμβάσει όπου αν είναι κάποιος ε, μεμονωμένος δικαιοδόχος, μπορεί να πάρει ε, καλύτερες τιμές από μόνος του αν ε, αντί να είναι μέλος ε, μιας ομάδας ας πούμε 30-40 επιχειρήσεων. Ως μικρός επιχειρηματίας μπορεί να έχει καλύτερα πλεονεκτήματα. Και το βασικό πρόβλημα σήμερα είναι ο ανταγωνισμός που δεν αγοράζει την, από τους δικαιοπαρόχους, τους δικαιοδόχους και βεβαίως η ψηφιοποίηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το βασικό πρόβλημα που εμείς θεωρούμε είναι ότι προκύπτει από τον ε, κανονισμό, ειδικά για τη ρήτρα για, την, ε, μη, για τον μη ανταγωνισμό, για τον κανονισμό 1330, ε, γιατί προβλέφθηκε για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό. Δεν ενισχύει τον ανταγωνισμό όμως, κατά τη δική μας άποψη, τον περιορίζει μάλιστα δείτε τον τίτλο. Μη ανταγωνισμός. Ρήτρα μη ανταγωνισμό. Εξαιρείται λοιπόν ο ανταγωνισμός. Οπότε υπάρχει αυτή η ρήτρα μη ανταγωνισμού στο τέλος της σύμβασής σας. Εμείς θέλουμε να περιορίζετε στην διάρκεια της σύμβασης. Φανταστείτε, έχετε μια επιχείρηση και σε ένα χρόνο πρέπει να κλείσετε την επιχείρησή σας ως αυτοαπασχολούμενο άτομο. Είναι ανταγωνισμός αυτό? Όχι βέβαια. Και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι δικαιοπάροχοι δεν θέλουν ο δικαιοδόχος να πάει σε, άλλη, σε άλλο όμιλο. Περιορισμός λοιπόν του ανταγωνισμού. Ο κανονισμός λοιπόν, ο 330, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό που ήθελε αρχικά να πετύχει. Επίσης, ο ορισμός της τεχνογνωσίας στον κανονισμό είναι πολύ ε, ασαφής. Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Ας πέρασω λοιπόν στα συμπεράσματα. Αυτορύθμιση. Είναι λύση? Όχι. Ο 72-2016 ε, δεν δίνει απάντηση στα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι κάθε μέρα. Και επίσης ε, δίνεται σημασία στο, στην ε, τεχνογνωσία. Η κωδική είναι α, μονομερής δεν δίνεται σημασία λοιπόν στους ε, δικαιοδόχους και επίσης ε, χάνεται πολύ χρόνο στην ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων για νέους κώδικες. Αυτό δεν είναι επιλογή για μας. Μία επιλογή ήταν να βελτιωθεί το σύστημα καταγγελιών. Ούτε αυτό λειτουργεί οι καταγγελίε είναι γνωστέ, τα παράπονα είναι σωστά. Και αν πάει κάποιο να παραπονεθεί ή να καταγγείλει, θα μπέσει, θα μπέσει στη ρήτρα τη μη δημοσίευση. Οπότε πάλι δεν του επιτρέπεται σε εισαγωγικά να καταγγείλει. Αυτοαξιολόγηση, ναι, το έχουμε αυτό ω οργάνωση. Υπάρχει δυνατότητα και μέσα αυτό, ε, για τους ε, ε, επιχειρηματίες για να αναλύσουν τη σύμβασή τους, αλλά όταν έχει συναυθεί η σύμβαση δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να την αναδιαπραγματευτεί. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ε, σαφές. το 330-2010 πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα, αλλά δεν θα λύσει τα άμεσα προβλήματα των δικαιοδόχων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να προσαρμοστεί, να τροποποιηθεί ο κανονισμός αυτός για να επιτύχουμε μια γενική λύση και για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην ψηφιακή εποχή. Ίσως να μπορεί αυτό να μπει στο refit. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν μέσω του refit να λύσουμε το πρόβλημα. Και επίσης καλύτερη ισορροπία στην εκπροσώπηση. Ναι βεβαίως, αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό και να υπερασπιζόμαστε φυσικά τα συμφέροντα των δικαιοδόχων. Θα σταματήσω εδώ και ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο που μου δόθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. And, uh, after the... Ευχαριστώ. Μετά από την έρευνα που ακούσαμε στις ε, Ολλανδικές πρακτικές και τις πρακτικές ε, στους, ε, στο χώρο των δικαιοδόχων, ας στραφούμε τώρα στους δικαιοπαρόχους. Έχουμε μια διπλή εκπροσώπηση. Έχουμε την κυρία Κάρολ Τσόπρα, που είναι η εκκριστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δικαιοχρησίας και την συνάδελφό της Νίκολα Βρότα. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, Ευχαριστούμε τον Ντένις Τεγιάν για τη δυνατότητα που μας δίνει να μιλήσουμε εδώ σήμερα. Μας παρουσιάσανε ως δικαιοπαρόχους. Αυτή, α, αυτό το κομμάτι της εξίσωσης. Αλλά είμαστε εδώ μια αντιπροσωπεία νέα ανθρώπων εδώ. Που είναι και δικαιοπάροχοι, που ξεκίνησαν την επιχείρησή τους στη δικαιοχρησία και ξεκίνησαν ως δικαιοδόχοι. Είναι εδώ επίσης νομικοί εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν είτε δικαιοπαρόχους, είτε δικαιοδόχους, είτε και τα δύο. Και με τους διευθυντές δύο ενώσεων της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας α, οργανώσεων δικαιοχρησίας. Ενθαρρύνουμε λοιπόν το κοινό να θέσει οποιαδήποτε ευαίσθητα ερωτήματα έχει για τις σχέσεις στη δικαιοχρησία και τη συμβάσεις δικαιοχρησίας στους ανθρώπους που είναι εδώ και που έχουν ζήσει όλα αυτά που ακούτε να παρουσιάζονται σήμερα. Θα εκφράσουμε τη θέση μας φυσικά. Όμως δεν εκπροσωπούμε είτε τους δικαιοπαρόχους είτε τους δικαιοδόχους ε, κάθε, και δεν βάζουμε κάθε τους φραγμούς ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. Ε, θέλουμε να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και οι αυτορυθμιστικοί κωδικοί εξυπηρετούν και τους δύο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικαιοχρησίας έχει το δικό της κωδικό για τους δικαιοπαρόχους. Υπάρχουν ε, αντίγραφα, μπορείτε να τα πάρετε καθώς θα φεύγετε και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή της Ολλανδίας να ετοιμάσει το δικό της κώδικα διοντολογία και νομίζω ότι πολλά πρέπει να γίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η παρουσίαση είναι εννιά διαφάνειες και θα παρουσιαστούν παράλληλα, ή μάλλον θα τις παρουσιάσω και εγώ και ο Νίκολα, που είναι από το, ή, Νίκολα, είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ε, επικεφαλής της ομάδας δικαιοχρησίας ε, στο νομικό της γραφείο και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Δικαιοχρησίας. Διάφοροι επισκέπτες μας είπαν ότι τους ενδιαφέρει η δικαιοχρησία. Ο στόχος μου λοιπόν καταρχήν είναι να σας πω ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε. Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί το χώρο της δικαιοχρησίας στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να πω ότι εκπροσωπούμε τον κλάδο αυτό, με βάση κάποια πρότυπα και κάποιες ε, δεοντολογίες. Δεν είναι μια τυφλή εκπροσώπηση του κλάδου, λοιπόν. Είναι μια στοχευμένη εκπροσώπηση. Μιλάμε για τα συστήματα δικαιοχρησία συνολικά. Και συμπεριλαμβάνουμε και δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους εδώ. Προωθούμε τη δικαιοχρησία ως ε, επιχειρηματική στρατηγική. Δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε το ένα από τα δύο μέρη μόνος. Η επιχειρηματική στρατηγική τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι δικαιοπάροχοι που υπερασπιζόμαστε και εκπροσωπούμε αποτελούνται, έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Και θα σας υπενθυμίσω ποια είναι αυτά. Επαναλαμβάνω ότι δεν εκπροσωπούμε αποκλειστικά τους μεν τους δε και ούτως ή άλλως λειτουργούμε με βάση κάποια πρότυπα. Και τον κλάδο της δικαιοχρησίας που δεν τα σέβεται δεν τον εκπροσωπούμε. Η δικαιοχρησία είναι ε, μια σύμβαση ανάμεσα σε δύο ανεξάρτητους επιχειρηματίες, σύμβαση B2B, όπου ένας δικαιοπαραχο ε, κάνει μια επιχειρηματική πρόταση σε έναν αγοραστή, ε, ο οποίος συμφωνεί να λειτουργήσει το σύστημα όπως ακριβώς ορίζει η σύμβαση. Πέραν αυτού, η δικαιοχρησία θα πρέπει να έχει τα εξή στοιχεία. Όλα. Χωρίς αυτά δεν θεωρούμε ότι η επιχειρηματική πρακτική είναι δικαιοχρησία. Που είναι ένα εμπορικό όνομα, ε, ε τεχνογνωσία και βοήθεια καθ' τη διάρκεια της σύμβαση. Τα IPR επίσης προστατεύουν τα στοιχεία του επιχειρηματικού πακέτου και γι' αυτό ο δικαιοπάραχος έχει το δικαίωμα να πάρει μέτρα ούτως ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα του εμπορικού σήματο, του δικτύου, ο δικαιοπάροχος δεν ασχολείται με έναν δικαιοδόχο και μόνο, αλλά με ένα δίκτυο ε, δικαιοδόχων, ε, εξού και η τυποποίηση, ας πούμε, των συμβάσεων δικαιοχρησίας. Ε, τεχνογνωσία. Ε, δεν, έχει δεν υπάρχει δικαιοχρησία χωρίς τεχνογνωσία. Ακούσαμε και ξέρουμε ότι η ύπαρξη της τεχνογνωσίας της συμβάσης δικαιοδοσίας αμφισβητείται και σε πολλές περιπτώσεις δικαίως. Η θέση μας είναι να πούμε ότι είναι καθήκον του δικαιοπαρόχου να ασχοληθεί με την τεχνογνωσία, πρέπει να επενδύσει, να αναπτύξει αυτή την τεχνογνωσία καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ε, είναι παρόν ούτω ώστε να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα στο εμπορικό σήμα και να βοηθήσει τον δικαιοδόχο να πουλήσει οτιδήποτε ας πούμε πρόκειται να πουλήσει και γι' αυτό είπαμε ότι ε, προωθούμε και υπερασπιζόμαστε τον, το know-how, την ε, τεχνογνωσία υπ' αυτή την ε, έννοια. Η Ομοσπονδία μας δεν ε, εκπροσωπεί μόνο αυτή την, αυτό το όραμα της δικαιοχρησίας, αλλά εκπροσωπεί και προωθεί και την αυτορύθμιση. Είμαστε πολύ υπέρ τη αυτορύθμιση, γιατί είναι ο καλύτερο τρόπο για να ρυθμιστούν οι σχέσει ανάμεσα στα δύο μέρη, δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Και ο κώδικα μα το επιβεβαιώνει. Μόλι θα αναθεωρήσαμε μάλιστα, η εκδοχή που είναι στη διάθεσή σα, λοιπόν είναι η τελευταία εκδοχή του κώδικά μα. Θα επανέλθω όμω στον κώδικα, στη τελευταία διαφάνεια και εδώ δεν θα πω άλλε λεπτομέρειε. Ένα τελευταίο σχόλιο για την Ομοσπονδία ε, Δικαιοχρησίας. Είμαστε μέλη, δεν έχουμε άμεσα μέλη εταιρείε, αλλά έχουμε ενώσεις ε, δικαιοδοσίας, όπου το δουσού τους έχει εκπροσώπους ε, δικαιοδόχων. Και πιστεύουμε ότι η καλύτερη πλατφόρμα για να προωθηθεί η δικαιοχρησία με τα πρότυπά της, τι αξίες κτλ. είναι να συνεργάζονται οι δικαιοπάροχοι και οι δικαιοδόχοι σε μια κοινή πλατφόρμα. Και καλωσορίζουμε την ε, εμπειρία των Ολλανδών που προσπαθούν να φέρουν κοντά τα δύο μέρη αυτά, ούτω ώστε να προωθηθεί ο κώδικας μέσω μιας κοινή πλατφόρμας. Θα δώσω τώρα το μικρόφωνο στη συναδελφό μου. Ευχαριστώ, Κάρολ. Καλησπέρα σα Όπως βλέπετε, η δικαιοδοσία ως ε, ε, επιχειρηματική στρατηγική είναι πολύ επιτυχής, ε, γεννά πολύ χρήμα σε πολλά κράτη-μέλη, πολλές θέσεις απασχόλησης και όλα, όπως όλα τα επιχειρηματικά συστήματα προσελκύει και καλούς και μέτρους και κακούς. Και δυστυχώ οι κακοί είναι αυτοί που του δίνουν το κακό όνομα. Αλλά δεν θα πρέπει όμω να αμαυρώνεται συνολικά η δικαιοχρησία, γιατί είναι πολύ πίκυλο πράγμα. Καλύπτει Πολλού τομεί αγορά, πολλού πολλούς διαφορετικούς κλάδους, είναι πάρα πολύ πολυπίκυλη ε, και υπάρχουν διαφορετικές συμφωνίες δικαιοχρησία. Και με ενδιαφέρον άκουσα τους εκπροσώπους του Ολλανδικού Υπουργείου να λένε ότι είναι κατά της ε, ενός μοντέλου σύμβασης ε, ντε και καλά. Γιατί η δικαιοχρησία είναι κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό και δεν υπάρχει μία σύμβαση που καλύπτει όλα τα είδη δικαιοχρησία. Θα πρέπει να προσαρμοστεί λοιπόν ανάλογα με το κράτο μέλο και τον κλάδο. Είναι οι δικαιοδόχοι, είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίε, δεν είναι καταναλωτέ, το είπε η μελέτη και θα πρέπει να έχει τον ίδιο βαθμό προστασία που έχουν οι καταναλωτέ στο δίκαιο ανταγωνισμού. Οι ανεξάρτητοι άνθρωποι μπορούν να ε, λάβουν νομικές συμβουλές, δέους επιμέλεια κτλ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δικαιοπάροχοι δεν δίνουν όλα τα στοιχεία στους δικαιοδόχους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δικαιοδόχοι δεν έχουν την υποχρέωση στη δέουσα επιμέλεια. Και αυτό το επιβεβαιώνουν και τα εθνικά δικαστήρια. Οι δικαιοπάροχοι επίσης είναι ΜΜΕ. Γενικά υπάρχουν μία-δύο μεγάλες εταιρείες ε, αλλά γενικά είναι με μία έψιλον ε. και θα πρέπει ε, να το έχουμε υπόψη μας όταν σκεφτόμαστε αν χρειαζόμαστε κάποιον νέο κανονισμό. Επίσης, ε, οι δικαιοπάρχοι εξαρτώνται από τους δικαιοδόχους για να επιτύχει η επιχείρησή τους. Είναι μια αμοιβαία σχέση. Εάν εκμεταλλεύεσαι μακροχρόνια το δικαιοδόχο, δεν θα επιβιώσεις. Η θέση της Ομοσπονδία μου είναι η εξή. Ότι η κάθετη φραγμή είναι απαραίτητη. Είναι υπέρ του ανταγωνισμού. Ε, με, στενή, με τη στενή, ο κανονισμός ε, μαζικών εξαιρέσεων έχει δίνει καθεντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις και λέει σε ποιες περιπτώσεις αυτή η φραγμή είναι αποδεκτή. Ε, στην πραγματικότητα βάζουν όμως κατόφλια στην αγορά ε, και προσπαθούν να μην ε, δημιουργήσουν καταχρήσεις. Ε, οι κανόνες των εθνικών δικαστηρίων είναι να εφαρμόσουν και να ερμηνεύσουν το δίκαιο του αγωνισμού για να αποφασίσουν σε ποιες περιπτώσεις, ε, οι κάθετε ή αυτοί φραγμοί έχουν τύχει ή ή μπορει να εφαρμοστούν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο δικαστηρίων των κρατών μελών. Οι κάθετοι περιορισμοί δεν είναι εγενείς α, αθέμητες πρακτικές. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούνται και άμα χρησιμοποιηθούν κακώς θα οδηγήσουν και θα γίνουν ε, κακές πρακτικές. Και αυτό ε, αναφέρθηκε και στον κανονισμό του 2003, α, τον 1200 και στα έγγραφα του Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια οριοθέτηση ανάμεσα στους κάθετους α, α, φραγμούς και στις ε, αθέμητες πρακτικές, αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τις αθέμητες πρακτικές δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε ε, ως ένα γενικό πράγμα που το χρησιμοποιούμε για όλες τις δικαιοχρησίες. Ε, αυτές οι πρακτικές ε, που, προσδιορίστηκαν στον τομέα των ε, τροφίμων έχουν ρυθμιστεί μέσω ε, αυτορύθμισης ή σε επίπεδο δικαστηρίων και δεν έχει ρυθμιστεί μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι να τροποποιήσουμε τον ανταγωνισμό μαζικών εξαιρέσεων δεν είναι η λύση στα προβλήματα της δικαιοχρησίας και δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο που ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, που έχουμε για να χρησιμοποιήσουμε. Ίσως υπάρχουν αθέμητες ρήτρε ε, σε συμβάσεις δικαιοχρησίας, αυτό λέει και η έκθεση, έχουν δοθεί μέσω παραδειγμάτων που δίνουν οι ίδιοι οι δικαιοδόχοι, προβλήματα που δεν βλέπαμε στην αρχή. Δεν θεωρούμε ότι η μελέτη ε, εκφράζει σωστά όλες τις πρακτικές των δικαιοπαρόχων σε όλη την ε, Ευρώπη. Εξάλλου, στον Ευρωπαϊκό Βασίλειο έχουμε μια πολύ όρημη αγορά, ας πούμε, δικαιοχρησίας. Τα παραδείγματα είναι ρήτρα μετά τον τερματισμό της σύμβασης ε, ε, ο δικαιοπάροχος ε, δεν είναι έτοιμος να δώσει τα εμπορικά του μυστικά ή τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα μάλιστα, θα πρέπει να προστατεύσει μάλλον την τεχνογνωσία του ε, και τα εμπορικά του μυστικά για να μπορέσει να διασφαλίσει την ε, επιχείρησή του. Ε, αυτή δηλαδή η διαφύλαξη του ε, εμπορικού μυστικού είναι σωστό να, γίνει, να υπάρχει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ε, επίσης, υπάρχουν αθέμητες πρακτικές των δικαιοπαρόχων όταν τελειώνει, τελειώνει τη σύμβαση ε, ο άμεσος ανταγωνισμός δημιουργεί προβλήματα. Ε, υπάρχουν κάποιοι δικαιοπάροχοι ε, που θέλουν να υποσκάψουν τη θέση των δικαιοδόχων πουλώντας το ίντερνετ, αλλά οι περισσότεροι ε, δικαιοπάροχοι ε, είναι σωστοί άνθρωποι, τίμοι κτλ. και μοιράζονται τις πληροφορίες τους ε, και μιλάνε για τις μεθόδους τους με τον δικαιοδόχο. Επίσης υπάρχουν κάποια κριτήρια επιδόσεων. Ε, συνήθως ε, υπάρχει αποκλειστικότητα όταν ο δικαιοπάροχος δίνει αποκλειστικότητα στον δικαιοδόχο. Ε, θα πρέπει να τον ελέγχει σε κάποιο βαθμό, γιατί δεν θέλεις να έχεις ένα μόνο δικαιοδόχο, ε, ο οποίος πάει τόσο χάλια, ας πούμε, ο οποίος θα σε θάψει. Ε, αυτό είναι σωστό, ε, φτάνει να γίνεται μέσα σε σωστά πλαίσια, μέσα σε σωστό ε, χρονικό διάστημα κτλ. Επίσης, ε, υπάρχουν κάποιες επικίνδυνες μεθοδολογίες. Ε, τα περισσότερα συστήματα ε, όμως είναι, δικαιοχρησίας είναι πολύ μικρά για να αντιμετωπιστούν από το δίκαιο ανταγωνισμού. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι ο δικαιοπάροχος ε, είναι ο κακός, ε, ότι είναι ο νικητής και ο άλλος είναι ο ιτημένος. Ε, και νομίζουμε ότι αυτή η γλώσσα δεν βοηθάει. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κάρδο για να σας πει τα καταληκτικά και να σας πει ποιες είναι οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για να διορθωθούν τα προβλήματα. Τα slides αυτά και όσα θα σας πω σχετικά είναι ακριβώς η ουσία των συμπερασμάτων μας, τα οποία λοιπόν θα διατρέξω. Όπως βλέπετε, είμαστε πολύ ευαίσθητοι στα θέματα που έχουν τεθεί από τις ενώσεις των δικαιοδόχων και των καταναλωτών. Είμαστε εκπρόσωποι του συνόλου των μικρομεσαίων τρόπων και είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών για να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς το όλο θέμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να προωθηθούν οι ανάγκες των μεν και των δε. Ω προ τα ενδίκα μέσα που συστήνει η έκθεση, αυτό που εμεί μπορούμε να πούμε, γιατί διαφωνούμε ελαφρώ, είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ω προ τον δίκαιο ανταγωνισμό. δεν νομίζουμε ότι. Δεν συμφωνούμε ότι αρμόζει, τέλο πάντων είναι η καλύτερη στρατηγική απλώς να προσαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την εξαίρεση 330 πριν από το 2022. Διότι ξέρουμε ότι από το 2022 θα καταργηθεί σιγά σιγά οποιοδήποτε σύστημα ε, διατομεακών περιορισμών στο δίκαιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι έχουν τη θέση τους ε, στο όλο αυτό το σύστημα, πρέπει απλώς να τις κατανοήσουμε καλύτερα και η έκθεση δεν εξετάζει με δίκαιο τρόπο όλη την ε, σχετική βιβλιογραφία που εξηγεί το πώς εφαρμόστηκε ως τώρα αυτή η εξαίρεση. Και η έκθεση καταλήγει σε μη σκόπιμες συστάσεις για τα ένδικα μέσα. Ως προς το ε, ευρωπαϊκό μέσο ε, επίλυσης διαφορών, αυτό το αμφισβητούμε. Ε, υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι αναφέρονται κατά λεπτό στα συμπεράσματά μας. Και όπως είπε και η Νίκολα, όταν τα ζητήματα ανταγωνισμού προκύπτουν σε συμβάσεις ε, δίκαιο χρυσίας, ακόμη και ζητήματα δικαίου και αδίκου, οι εθνικές νομοθεσίες αρκούν. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν ε, την σχετική αρμοδιότητα από τον κανονισμό του 2003 και, τα ευρωπαϊκά, και οι νομικές υπηρεσίες είναι αρκετά καλά εξοπλισμένες για να ενημερώσουν για τα ενδικά μέσα που προσφέρονται στους εμπορευομένους. Όπως είπα, η Ομοσπονδία μας ε, πιστεύει κράδαντα ότι η αυτορύθμιση πρέπει να επικρατήσει και ο κώδικας που σας διατίθεται θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά και την εξέλιξη του ραντικού κώδικα. Ας προ την εκπροσώπηση, το θέμα της ε, άδικης εκπροσώπησης ότι υποεκπροσωπούνται μάλλον οι δικαιοδόχοι, το έχω πει εδώ. Έχουμε επιχειρηματίες που ήταν, που ήταν δικαιοπάροχοι και μετά έγιναν δικαιοδόχοι. Δυσκολεύονται οι δικαιοδόχοι δύσκολα ε, καταφέρουν να παρίστανται στις πλατφόρμες συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών. Διότι είναι αποσχολημένοι με την ε, οργάνωση των επιχειρήσεών τους. Όμως πιστεύουμε ότι οι πλατφόρμες αυτές εκπροσωπούν και τους δύο. Και μια κουβέντα για τον δικό μας κώδικα και το μηχανισμό, με συγχωρείτε, αλλά έχετε πάρει το διπλάσιο χρόνο σε από αυτό που σας αναλογούσα και δεν θα προλάβουμε. Έχω μια πολύ γρήγορη ερώτηση που ίσως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και στα αντεπιχειρήματά σα. Λέτε ότι μπορείτε να, μπορεί να επηρεαστεί ο Ελλανδικό κώδικα, ότι να γίνει πολλή δουλειά προ αυτό. Όμω, η ε, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων μα είπε ότι αυτό είναι ο κώδικα. Δεν φαίνεται να έχει ανάγκη από περαιτέρω δουλειά. Τι δουλειά εντοπίζετε εσεί ότι χρειάζεται, τι διόρθωση, ποια είναι τα σημεία στα οποία διαφωνείτε με τον κώδικα. Δεν διαφωνώ. Απλώ θα θέλαμε το πνεύμα και το κλίμα του οποίου γίνονται οι διαπραγματεύσει να εκφράσει την πλήρη συνεργασία, εμπιστοσύνη και διάθεση να προχωρήσουμε μεταξύ των δύο πλευρών. Είστε υπέρ αυτού του πνεύματο και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε και από τη συνένεση στην οποία καταλήξαμε ο κώδικα. Και τώρα θα ακούσουμε τον δόκτωρα Μάρκ Άμπελ, ο οποίο είναι πραγματικά εμπειρογνώμων για την ε, αδειοδότηση των ε, δικαιοδόχων έχει εργαστεί σε νομική εταιρεία, την Bird and Bird, και επίσης ε, στον ύπρο τον ε, Διεθνή Οργανισμό για την Θεματική Ιδιοκτησία και σε πολλούς εμπορικούς οργανισμούς. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα και αν μπορείτε να περιοριστείτε λιγάκι στο χρόνο σα σας για να έχουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επί 35 χρόνια, επί καθημερινής βάσης, ως ακαδημαϊκός και ε, νομικός, έχω ασχοληθεί με την δικαιοχρησία, δίνοντας συμβουλές και σε δικαιοπαρόχους και σε δικαιοδόχους. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω αρκετό χρόνο για να διατρέξω τα πάντα που έχουν σχέση με τι δικαιοχρησίε και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα. Θα σα δώσω λοιπόν μόνο κάποιες ε, τηλεγραφικές παρατηρήσεις. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες που θα ήθελα να σα παρουσιάσω, αλλά τρία είναι τα βασικά γεγονότα στα οποία θέλω να σταθώ. Πρώτον, η δικαιοχρησία δεν δίνει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτυγχάνει αυτά που επιτυγχάνει σε άλλες οικονομίες, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, οπουδήποτε. Οι επιδόσεις της είναι χαμηλότερες. Αυτό θα πει ότι ως οικονομική αγορά δεν αποκομίζουμε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη. Δεύτερον, αυτές οι χαμηλότερες επιδόσεις σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ρυθμίζεται το σύστημα των δικαιοχρησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κάτι μελη έχουν ε, ορίσει διαφορετικούς κανόνες και συστήματα κανόνων για τη δικαιοχρησία και ε, αν τα προσθέσει κανείς δημιουργούν τεχνικούς φραγμούς ε, στην εξάσκηση και την υλοποίηση της δικαιοχρησίας που δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικαιοχρησία επικεντρώνεται σε μικρό αριθμό των ευρωπαϊκών κρατών Τρίτο στοιχείο. Προκειμένου να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά, πρέπει όλος χερός να αναθεωρήσουμε το σύστημα των κανόνων. Όπως τα λέγει ο Σον πατών, να δημιουργήσουμε έναν αντιπερισπασμό. Μια διαφορετική προσέγγιση δηλαδή. Ε, ακούσατε κάποιες αναλύσεις που ήταν αρκετά ε, ριζικές. Ε, και η καθεμιά υπερασπιζόταν διαφορετική άποψη. Με κάποιες συμφωνώ, με κάποιες όχι από τις παρατηρήσεις που ακούσαμε. Πάντως, οι δικαιοδόχοι δεν είναι πάντοτε αθώοι και αφελής. Ε, μερικές φορές ναι, μερικές όχι. Κάποιες φορές είναι και μεγαλύτεροι και πιο ισχυροί από τους δικαιοπαρόχους τους. Και αυτό δεν ισχύει πάντοτε, αλλά είναι γεγονός. Δεν είναι πάντως μια διμερής σχέση. Ο δικαιοπάροχος σε τοπικό επίπεδο πρέπει να συμπεριφερθεί έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι δικαιοδόχοι σε όλη την αλυσίδα της συνεργασίας τους ε, είναι, έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και δεν ε, δίνει ατομικά σε κάθε δικαιοδόχο ξεχωριστή μεταχείριση. Είναι αρκετά πολύπλοκο το σύστημα. Να δούμε πώς μπορεί αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι κάπως κάνω άλματα μεταξύ των διαφανειών μου, διότι θα ήμασταν εδώ για πολλές ώρες αν έπρεπε να αναλύσω όλα. Για πάμε λίγο πίσω. Αυτορύθμιση. Ακούσαμε πολλά για την αυτορύθμιση. Έχω περάσει πέντε ολόκληρα χρόνια ε, αναλύοντας το εάν δουλεύει και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι όχι. Η αυτορύθμιση δεν δουλεύει. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο τη Ομοσπονδία Ευρωπαϊκή Δικαιοχρησία και των σχετικών ενώσεων, αλλά μην αυταπατώματα. Η δικαιοχρησία δεν μπορεί να ρυθμιστεί επιτυχώ, κατά την άποψή μου, με την ε, βάση της ε, αυτορύθμιση τη απολύτω ελεύθερη. Εάν αναλύσει κανείς τον τρόπο που οι ενώσεις δικαιοχρησίας προσπαθούν να αυτορυθμιστούν με την πάροδο των ετών, βλέπει ότι δεν είναι και πολύ επιτυχής ο τρόπος τους. Η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έφερε πολλές θετικέ συμβολέ στη δικαιοχρησία, πρόθυσαν κάποια πράγματα και μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερο, όμω η αυτορύθμιση από μόνη τη δεν θα είναι η λύση. Τρία βασικά εμπορικά στοιχεία πρέπει επιτακτικώ να ισχύσουν και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Η δικαιοχρησία μπορεί να είναι ένα δώρο, μια ευλογία για την ευρωπαϊκή οικονομία, εάν την εκμεταλλευτούμε στο πλήρε δυναμικό. Πρώτον, πρέπει να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς στη δικαιοχρησία. Για πάμε λίγο πιο πέρα, ναι, σε όλο αυτό το κεφάλαιο. Ε, Πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Εάν πραγματικώς επιτύχει η δικαιοχρησία, πρέπει να προσελκύει επιχειρήσεις που θα την χρησιμοποιούν ως τρόπο να ε, βελτιώσουν τις δραστηριότητες τους. Δηλαδή, να μην είναι απλώς ραβδί ο κανονισμό και το σύστημα των κανόνων μας να μην είναι τιμωρητικός, να μην λέει απλώς τους ε, δικαιοδόχους τι πρέπει να κάνουν, να υπάρχει μια ανταλλαγή, να υπάρχουν ωφέλη, να υπάρχει κάτι που προκύπτει για τους δικαιοπαρόχους. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει κανείς να εμπορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο, αν υπεριθμίσει κανείς την δικαιοχρησία αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα το ονομάσουν αλλιώ οι άνθρωποι, θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο που κάνανε πριν, αλλά θα περιεφηρεοποιηθεί το συγκεκριμένο σύστημα. Δηλαδή θα αποκλειστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κατά τα άλλα θα διαδοθεί περισσότερο. Α ενθαρρύνουμε λοιπόν τι επιχειρήσει να καλλιεργούν την δικαιοχρησία, να τη χρησιμοποιούν, βλέποντα όμω χειροπιαστά ωφέλη ε, από το να είναι, γίνεται κανεί δικαιοπάροχο. Δηλαδή μαζί με το ραβδί να χρησιμοποιούμε και το καρότο. Ε, εάν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς, θα είχα πολλά να προτείνω και θα δώσω κάποια παραδείγματα πολύ γρήγορα. Λόγου χάρη, οι δικαιοπάροχοι θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν από τους δικαιοδόχους να αποκαλύπτουν όλα τους τα στοιχεία πρώτης υπογραφής της συμβάσεως, όπως και οι ίδιοι. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτει στι διαδικασίε επίλυση διαφορά από τα 35 χρόνια μου εμπειρία στην δικαιοχρησία δεν είναι οι κακοί δικαιοπάροχοι, ούτε οι κακοί και τεμπέληδε δικαιοδόχοι. Είναι το εξή, ότι δεν γίνεται σωστή αντιστοίχηση των προσδοκιών των ΜΑΡ και των δε. Δηλαδή, ο δικαιοπάροχο και ο δικαιοδόχο δεν ε, κατανοούν πλήρω τη σχέση στην οποία, ε, την οποία εκκινούν με τη σύμβαση. Πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Εάν πρόκειται να ρυθμίσουμε τη δικαιοχρησία, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι επικεντρωνόμαστε στα τμήματα εκείνα τη δικαιοχρησία που μπορεί να είναι αποφελή. Δηλαδή να αποκλείσουμε μικρού ε, δικαιοπαροχού, αυτούς που μπορεί να είναι μόνο κλασματικοί, αυτούς που μπορεί να είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι, τεράστιοι ή αυτοί που μπορεί να έχουν ε, ε, Πληροφορίε εκ των έσω. Να ρυθμίσουμε αυτού που χρειάζονται ρύθμιση. Αυτό που πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι οι αλυσίδε δικαιοχρησίας μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ ε, σε σχέση με μεγάλους ομίλου. Υπάρχει άποψη ότι πολλά από τις ε, μαζικές εξαιρέσεις και οι υπόλοιποι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφελούν τους μεγάλους ε, οικονομικούς ομίλους και όχι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι στη θέση του δικαιοπαρόχου είτε του δικαιοδόχου. Γι' αυτό σε, μια, σε ένα νέο σύστημα κανόνων, αυτό που θα ήθελα να δω είναι οι δικαιοπάροχοι, όπως και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, να μπορούν να επιβάλλουν μια τιμή, ε, μια πολιτική τιμών γιατί αυτό θα στηρίξει την ε, προσπάθειά τους. Είναι η τιμή που είναι το θέλγητρο. Ε, θα ήθελα επίσης να υπάρχει ένα καλύτερος τρόπος να ελέγχουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται. Δεν νομίζω ότι ο δικαιοπάροχος θα έπρεπε να βρίσκεται σε σχέση ανταγωνισμό με τον δικαιοδόχο, όμως δεν θέλω και οι δικαιοδόχοι να έχουν το δικαίωμα να εξεγερθούν και να κάνουν στο διαδίκτυο ό,τι τους αρέσει με το σήμα του δικαιοπαρόχου. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει υγιεινή πρώτη υπόγραψη τη σύμβαση. Εδώ είναι το σημείο που οι προσδοκίε των ΜΕΝ και των ΔΕ δεν αντιστοιχούνται. Ε, είναι σημαντικό οι δικαιοδόχοι να ε, υποχρεούνται να ε, λάβουν τι απαραίτητε συμβουλέ πρωτού υπογράψουν τη σύμβαση. Δηλαδή να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το στάδιο και στι συμβουλέ που θα λάβουν και οι συμβουλέ να προέρχονται από νομικού και λογιστέ που πραγματικά κατανοούν, κατανοούν τι πρόταση έρχεται στα χέρια τους. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουν να διαδραματίσουν οι εθνικές ενώσεις ε, των δικαιοδόχων. Θα πρέπει να διευκολύνουν την κατανόηση και να βεβαιωθούν ότι οι νομικοί που παράσχουν συμβουλές τους ε, δικαιοδόχους γνωρίζουν κάποια πράγματα για την δικαιοφρυσία ότι έχουν περάσει ένα μάθημα στο διαδίκτυο λόγω χάρη, μια εκπαίδευση. Αλλά οι δικαιοδόχοι πρωτού υπογράψουν θα πρέπει πραγματικά να έχουν ε, δώσει πιστοποιητικό από έμπειρο νομικό ε, με μακρά εμπειρία στις συμβουλές για το δικαιοχρησία λέγοντας ότι όντως κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Οι δικαιοδόχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να ε, παρακολουθήσουν και αυτοί ένα βασικό μάθημα για το τι είναι η δικαιοχρησία και τι απαιτήσει θα αναλάβουν να εκπληρώσουν. Αυτά μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με ενώσεις δικαιοδοχών. Μπορεί εν μέρη να χρηματοδοτηθούν αυτά από ευρωπαϊκά κονδύλια ή τις εθνικές κυβερνήσεις και θα πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν στη δικαιοχρησία ε, το τι αναμένεται από αυτούς. Να το ε, καλλιεργήσουμε αυτό. Έτσι θα καταλάβουν τι σημαίνει η αποκάλυψη πληροφοριών πρώτη υπογραφή τη σύμβαση. Μπορεί κανεί να δώσει πληροφορίε θέλει ω αλλά αν ο δικαιοδόχο τα διαβάζει και δεν τα καταλαβαίνει, δεν έχει νόημα. Οπότε αυτή η υγιεινή εντό εισαγωγικών πρώτη υπογραφή τη σύμβαση είναι σημαντική και θα πρέπει να ε, ισχύσει σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Προς στιγμήν έχουμε έξι διαφορετικές απαιτήσει, έξι διαφορετικά συστήματα περί απέτηση αποκάλυψης πληροφοριών, τα οποία είναι όλα διαφορετικά, είναι μεταξύ τους αντικρουόμενα και τελικά οδηγούν σε διαφορετικούς, ε, στην ε, δημιουργία διαφορετικών φραγμών, ώστε να μην μπορούν οι δικαιοπάροχοι να συνεργαστούν αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος πανευρωπαϊκός κώδικας. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με το να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφές το τι αναμένεται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή να υπάρχει μια σειρά από όρους ε, δεσμευτικούς σε όλες τις συμφωνίες δικαιοχρησίας και να καθίσταται σαφές τι πρέπει να πετύχει ο δικαιοπάροχος και τι πρέπει να κάνει ο δικαιοδόχος. Είναι ε, αλήθεια, αναντήρητη, ότι λάζουν οι υποχρεώσει των δικαιοπαρόχων από επιχειρήση σε επιχειρήση. Το ξέρω γιατί όλη τη μέρα, κάθε μέρα με αυτά ασχολούμαι. Αλλά ω νομικό που καθημερινά ασχολούμαι με αυτό το θέμα και ω ακαδημαϊκό που έχω ασχοληθεί πέντε χρόνια με τη σχετική έρευνα για να μελετήσω τα είδη συμφωνιών σε όλα τα κράτη-μέλη, ότι όλοι έχουν βασικές, βασικά κοινά στοιχεία. Αυτά τα κοινά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε συμφωνία. Δεν θα τα δω ε, κατά λεπτός, ποιες πρέπει να είναι αυτές οι διαφορετικές απαιτήσει, όμως, λόγω χάρη, ο δικαιοπάροχος έχει λόγω χάρη δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Οι δικαιοδόχοι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το αμφισβητήσουν. Οι δικαιοπάροχοι θα πρέπει να παρέχουν εξωπρεπή εκπαίδευση και να μην επιτρέπεται να ε, πιέσουν τους ε, δικαιοδόχους προσπαθούν να τους κλέψουν πελάτες. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Κι όμως η μεγάλη πλειοψηφία των ε, δικαιοπαράχων σήμερα από όσα έχω δει εγώ, δεν το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Οι δικαιοπάροχοι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη δικαιοχρησία σαν εφαλτήριο για να κερδίσουν πολύ περισσότερα στη δική τους επιχείρηση οι ε, δικαιοπάροχοι θα μπορούσαν να είναι μικρέ επιχειρήσει. Εάν ο δικαιοδόχο επίση μπορεί να κλέψει ε, την πνευματική διεκτησία ενό δικαιοπαρόχου και να τη χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή επιχείρηση ω παρακλάδι, αυτό βεβαίω ε, είναι μια μορφή του να ε, μην αντιδρούμε μπροστά στην απάτη, να την ε, αποδεχόμαστε. Η εμπιστευτικότητα. Ακούσαμε πολλά για το πώς οι δικαιοπάροχοι κερδίζουν χρήματα. Για το πώς πληρώνουν περισσότερα για κάποια πράγματα από ότι ανεξάρτητοι traders. Αυτό δεν έχει σχέση με την ουσία του θέματος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι δικαιοδόχοι γίνονται δικαιοδόχοι, πρέπει να ε, γνωρίζουν σαφώς πώς ο δικαιοπάροχος κερδίζει ε, χρήματα. Αυτό ε, ε, μπορεί να έχει να κάνει με τα προϊόντα, αλλά πρέπει να είναι σαφές, ξεκάθαρο και ανοιχτό. αυτό είναι βέβαια εμπορική απόφαση κατά την δική μου, από τη δική μου την εμπειρία. Πολύ συχνά. Ακόμη και αν κάποια από τα προϊόντα είναι ακριβότερα για τους, δικαιοδόχους και αυτό είναι τελείως ασυνήθιστο. Αλλά αν συμβεί ας πούμε, είναι πραγματικά αποτρεπτικό, εάν δει κανεί την ε, εικόνα του εμπορικού συστήματος συνολικά. Διότι κερδίζει περισσότερα χρήματα ο δικαιοπάραχος έτσι κι Εάν δείτε τι γίνεται στην Αυστραλία και τι ΗΠΑ, συνολικά το ποσοστό αποτυχία των μικρών επιχειρήσεων που δεν είναι δικαιοδόχοι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των δικαιοδόχων. αυτό δεν σημαίνει ότι οι δικαιοδόχοι δεν αποτυχάνουν. Κάποιε φορέ φτωχεύουν. Δεν είναι εγγύηση επιτυχία η μας είμαστε σαφεί. Είναι ένα αποτύπωμα, για να το πω έτσι, μια επιχείρηση. Είναι αποτύπωμα που ε, με τη δοκιμή και την πλάνη δημιουργείται και ενισχύεται και με την περίοδο του χρόνου. Αυτό το αποτύπωμα διατίθεται στους δικαιοδόχους και μπορούν να το αξιοποιήσουν. Δεν αποτελεί εγγύηση όμως. Εάν τα δούμε λοιπόν όλα αυτά μαζί, πού καταλήγουμε ότι ο τρόπος που τώρα έχουμε ρυθμισμένη την δικαιοχρησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως άσκοπος. Ε, δημιουργεί εσωτερικούς τεχνητού φραγμούς και δεν, ε, δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει όλα τα δυναμικό τη δικαιοχρωσία είτε από την πλευρά των δικαιοπαρόχων, είτε των δικαιοδόχων, είτε και των καταναλωτών. Και πραγματικά σα συστήνω να ακολουθήσετε την προσέγγιση της οδηγίας. Υπάρχει πρόταση ε, για τη σύνταξη της οδηγίας προς τον ε, πρόεδρο. Ε, μέρος του διδακτορικού μου ήταν αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο σκόπιμο μπορούμε να κάνουμε και αυτό θα πρέπει να κάνουν και οι Εθνικές Ενώσεις των Δικαιοπαρόχων, παρόλο που κάπως διαφέρει από την προσέγγιση στην οποία έχουμε για την ώρα εμπλακή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσουμε τις ε, διαφάνειές σας ε, για, ως πηγή έμπνευσης για, ε, για την έκθεση που ίσως συντάξουμε το καλοκαίρι. Έχουμε ξεπεράσει λιγάκι το, το χρόνο μας. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει στις 4.25 το πρώτο πάνελ και είναι ήδη 5 παρατέταρτο. Έχουμε μέχρι τις 5.30 μέσα σε τούτη την αίθουσα. Οπότε καλό θα ήταν να πάμε κατευθείαν στο επόμενο πάνελ και να ζητήσουμε από τους ομιλητές το επόμενο πάνελ να είναι πολύ σύντομοι έτσι ώστε στο τέλος να καταφέρουμε ίσως να, κάνουμε, να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τους επόμενους ομιλητές. Η κυρία Κριστέλ Ντελμπέργκε από το Eurocommerce, η Πατρίτσια Χόχστράτεν από το VAC Centrum και η δόκτωρο Ντάβια Βουένο να έρθουν εδώ στο βήμα για να τους ακούσουμε. The um, first member of this panel who will speak is uh, Christa Η κυρία Δελμπέργκε θα μας μιλήσει πρώτη. Είναι υπεύθυνη για την ανταγωνιστικότητα και τις ε, δημοσίευσει στην ε, Eurocommerce. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Τιγιόγκε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί νομίζω ότι πολλά από όσα είχα να πω ε, υπόθηκαν από τους ομιλητές του πρώτου πάνελ. Να πάμε στην αμέσως επόμενη διαφάνεια. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ έχει να κάνει με την σημασία του λιανεμπορίου στην δικαιοχρησία. Και βεβαίως θα περάσουμε στην, και στα κάποια συμπεράσματα και σε προτάσεις. Η Eurocommerce λοιπόν είναι μια ε, οργάνωση που εκπροσωπεί ομοσπονδίε ενώσει από 30 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Έχουμε μέλη σε όλα τα ευρωπαϊκά, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από δύο. Έχουμε ομοσπονδίε τομεακέ. και 30 ε, περίπου ε, ε, επιχειρήσεις ε, πρωτοπόρους στον, ε, στο λιανεμπόριο. 5,5 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο λιανεμπόριο. Απασχολούν 30 εκατομμύρια άτομα και έχουν 10% του ΑΕΠ. Μιλούμε για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και μεταποίηση το λιανεμπόριο και το χονδρομόριο κυριαρχείται από πλειοψηφία μικρών ε, επιχειρήσεων που, είναι το, που, απασχολούν το 2 τρίτο των απασχολούμενων και έχουν ένα ΑΕΠ 35%. Ε, ε, Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, στην, και στο λιανεμπόριο και στο χοντρεμπόριο είναι μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, δραστηριοποιούνται σε, μεγά, σε πολύ ανταγωνιστικό και συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον και βεβαίως πρέπει πάντα να ε, προωθούν την καινοτομία στην Ευρώπη και αντιμετωπίζουν σαφώς πάρα πολλές προκλήσεις όπως η ε, ε, μεταπίδηση στην ψηφιακή εποχή αλλά και η περίπλοκη νομοθεσία, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η διαθεσιμότητα της κατάρτισης του προσωπικού και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. Επίσης υπάρχουν διάφοροι όμιλοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να μπορούν να το σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, λίγα λόγια για να τονίσουμε την σημασία της δικαιοχρησίας, κυρίως στο δικό μας τομέα, αλλά γενικώ η δικαιοχρησία είναι πολύ σημαντικό μοντέλο επιχειρησιακό, δημιουργεί πραγματικά μεγάλη ε, ε ανάπτυξη και επίσης ε, θέσεις 500.000 outlets υπάρχουν στην Ευρώπη, 14.000 εμπορικά σήματα, πάνω από 3 εκατομμύρια απασχολούμενοι, εργαζόμενοι. Είναι ε, εύκολο ο τρόπο αυτό να έχει κανεί πρόσβαση στην αγορά και, να, και σε νέε αγορέ και για του δικαιοπαρόχου και για του διοδόχου. Οι δικαιοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να διαρευνήσουν τα ωφέλη και να έχουν νέε εμπορικέ φόρμουλε και να διαχειριστούν τι επιχειρήσει του ω επιχειρηματίε. Και επίση ο δικαιοπάροχο μπορεί να μπει σε νέε αγορέ και να εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία αλλά και την ε, δυνατότητα του ε, δικαιοδόχου να ε, διαχειριστεί εξ ονόματός του την φόρμουλα. Επίσης, βρίσκονται στις, σε πολύ μεγάλες πόλεις αλλά και σε πολύ μικρές πόλεις και σε εμπορικά κέντρα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και αυτό είναι πιο, καθιστά πιο εύκολη την διαχείριση της επιχείρησης από τους δικαιοδόχους και την εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη. Υποστηρεί, το, η δικαιοδοχία υποστηρίζει την κοινοτομία και την τεχνογνωσία που αλλιώς δεν θα ήταν ήταν προσβάσιμε σε ε, μεμονωμένου επιχειρηματίε, οπότε η δικαιοχρησία είναι πάρα πολύ σημαντικό επιχειρησιακό μοντέλο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ήθελα να πάμε λίγο να δούμε τον ορισμό της ε, ε αλλά νομίζω ακούσαμε πολλά σχετικά. Δύο σημαντικά στοιχεία όμως ε, σχετικά με τόσα υπόθηκαν. Η δικαιοχρησία δεν είναι λιανεμπόριο. Είναι μια φόρμουλα επιχειρησιακή που ε, ε, εμπλέκεται σε πάρα πολλούς ε, τομείς της οικονομίας. Οπότε θα ενθαρρύναμε όλους να έχουν μια ευρεία προσέγγιση όταν μιλούν για, το, για τη δικαιοχρησία, γιατί δεν είναι ένας τομέας στη δικαιοχρησία, είναι ένα μοντέλο. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι η ποικιλία των σχέσεων των δικαιοχρησίας και, των, και της φόρμουλας που υπάρχει. Είναι δύσκολο να βρούμε μια πανάκια για όλους, ε, γιατί υπάρχουν διαφορετικές υποχρεώσει από την πλευρά των ε, δικαιοδόχων για την ε, εκμετάλλευση της φόρμουλας και αυτό βεβαίω πρέπει να, αντιστοίχως πρέπει να, από την πλευρά των ε, δικαιοπαρόχων να γίνεται σεβαστό ε, το προϊόν τους. Πρέπει βεβαίως ο δικαιοδόχος να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ένα ποσοστό του, ε, του προϊόντος εκτός της δικαιοχρησίας. Θα υπάρχουν βεβαίως περιπτώσεις και έχουμε ακούσει πολλές όπου ο δικαιοπάροχος μπορεί να μην είναι το ισχυρό μέρος στην συμβατική σχέση. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση θέλει να μπει σε μια νέα εθνική αγορά, θα διαπραγματευτεί με έναν operator για να αναλάβει την δικαιοχρησία, τη σχετική άδεια για όλη την αγορά. Οπότε έχουμε, υπάρχουν όλων των ειδών οι ασυμμετρίες και οι διαφορετικών ειδών σχέσεις στην δικαιοχρησία. Οπότε δεν υπάρχει μόνο ένα είδους σχέση συμβατικής. Επιλογές πολιτικής. Εμείς θα ενθαρρύναμε ε, έντονα τους ε, Χαράζοντα την πολιτική να καθορίσουν λιγάκι τα δεδομένα. Η ε, διοχρησία χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία πληροφοριών και ε, δυσκολίες που δημιουργούνται από την ύπαρξη των μικρών παιχτών. Είναι πολύ περίπλοκη λοιπόν σχέση. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα και με την ατζέντα για την καλύτερη διαχείριση, πριν καταλήξουμε στα συμπεράσματα και πριν κάνουμε συστάσεις για την πολιτική, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα δεδομένα, να δούμε δηλαδή τις, ε, ε, τα, τα, τα ταλέντα που υπάρχουν στην αγορά και παρόλο που υπάρχουν κάποιες ε, υποθέσεις στα δικαστήρια, Μπορεί να υπάρχουν ε, θέματα εμπιστευτικότητα των ε, συμβάσεων. Ε, παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά πολλά προβλήματα έχουν αναφέρει οι ερευνητές, οι λύσεις για τα οποία όμως δεν αποτελούν όντως λύσεις ε, όπω είπα, η δικαιοσύνη είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο και δεν αφορά έναν ένα αποκλειστικό τομέα. Οπότε, αν υπάρχει ανάγκη για δράση, θα πρέπει να βασίζεται στην εξέταση του μοντέλου και να μην συνδέεται με, την, με συγκεκριμένη προσέγγιση. Η προτινόμενη λύση για την αναθεώρηση των, ε, του κανονισμού για, την, ε, για τι συνολικέ εξαιρέσει εξετάζει τι σχέσει με του δικαιοπαρόχου, τον ανταγωνισμό και του κανόνε ανταγωνισμού, η προστασία στην αγορά και το όφελο προ τον καταναλωτή. Δεν θέλουμε να ε, προστατεύσουμε μέρη ή μεμονωμένους τομείς μέσω διμερών σχέσεων. Η μεμονωμενου τομεί μεσω διμερων σχεσεων η δικαιοχρησια και οι σχέσεις τη καλύπτονται από το ιδιωτικό δίκαιο και τα σχετικά μέσα όπως η ε, δέουσα ε, δράση στην αγορά. Αυτό εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, αλλά έχει, στόχο τον, έχει τον ίδιο στόχο. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες, υπάρχουν εθνικοί κανόνες, υπάρχει το, το νομικό ε, περιβάλλον και κατά την άποψή μας το εθνικό επίπεδο είναι το καταλληλότερο για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Η αποτυχία να υιοθετηθεί ε, ένα κοινό ε, σχέδιο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει την δυσκολία να υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα του συμβατικού δικαίου ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέσα του ιδιωτικού δικαίου μπορεί να συμπληρωθούν από του κανόνε διοντολογία και η EFF έχει εκπονήσει έναν τέτοιον, καθώ επίση και εργαλεία με τη δυνατότητα να κωδικοποιηθούν οι κώδικε σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση από πολλού ε, παράγοντες ε, και από την ομάδα που δημιούργησε το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν δύο μέρη στο τραπέζι και εμείς ενθαρρύνουμε και, τους, και τις δύο πλευρές να, να δούνε τα μέσα αυτορύθμισης και πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στην εθνική τους κατάσταση. Συμπερασματικά λοιπόν ζητούμε μια προσεκτική προσέγγιση που θα βασίζεται στα δεδομένα γιατί μιλούμε για ένα επιχειρησιακό μοντέλο και όχι για ένα συγκεκριμένο τομέα και η προσέγγιση προ την δικαιοχρησία θα πρέπει να ε, αφορά στη σχέση και όχι στον τομέα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ε, επιλογή των ε, μέσων πολιτικής και η αυτορύθμιση θεωρούμε ότι είναι η Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε, Κρυστάλλου. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Πατρίσια Χολτ που είναι όχι μονογενική γραμματέας της Center, Είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Συμβουλίου στην Ολλανδία και μέλος της βασιλικής οργάνωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων γνωρίζει πάρα πολύ καλά την δικαιοχρησία. Πατρίσια, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους των Βέλγων και Ολλανδών δικαιοδόχων, ευχαριστώ την Επιτροπή ΙΜΚΟ για την μελέτη αυτή που παραγγείλατε. Παρατηρήσαμε ότι τα πορίσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις που κάναμε στο παρελθόν τα τελευταία δέκα χρόνια. Ότι καλές και πρακτικές λύσεις ε, δεν έχουν ακόμα βρεθεί. Και η κατάσταση χειροτερεύει από τη στιγμή που η δικαιοχρησία αναπτύσσεται ως πρακτική. Υπάρχει μια αίσθηση κατεπήγοντος. Η δικαιοχρησία ε, και τα μέλη των δικαιοδόχων ε, κάνουν έκκληση στις εθνικές γραμμές, στις εθνικές αρχές. Ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν σημεία επαφής και να συλλεχθούν περισσότερες ε, πληροφορίες μεν, που όμως δεν μπορεί από μόνες τους να υποστηρίξουν τους δύο δικαιοδόχους. Θα πρέπει πάρα αυτά να λάβετε τα απαραίτητα βήματα, ούτως ώστε να διασφαλίσετε το μέλλον των ανεξάρτητων επιχειρηματιών που συνεργάζονται ε, και δουλεύουν στα πλαίσια της δικαιοχρησίας. Δεν βλέπω τις διαφάνειές μου όμω στον πίνακα. Α, είναι στον έναν από πίσω μου μόνο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν οι φραγμοί στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο κανονισμός 330 αρχικά είχε σκοπό να εξασφαλίσει και τον ελεύθερο ανταγωνισμό καθώς και την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, εμείς ε, συμφωνούμε με το συμπράσμα της μελέτης ότι το δίκαιο ανταγωνισμού έτσι ως έχει δεν είναι λειτουργικό για τον τομέα της δικαιοχρησίας. Η θέση των δικαιοπαρόχων ενισχύεται περαιτέρω από τον κανονισμό αυτό. Και το ερώτημα που τίθεται στο κεφάλαιο 8 της μελέτης, το μοντέλο της δικαιοχρησίας είναι κατάλληλο ε, για τον κανονισμό αυτό, δείχνει ότι η μοντέρνα δικαιοχρησία ε, δεν ρυθμίζεται, ε, δεν εντάσσεται καλά στο πλαίσιο του καονισμού. Ε, δεν λάβαμε υπόψη στο ηλεκτρονικό εμπόριο ε, και διάφορα άλλα στοιχεία. Η δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει αναλογικότητα ανάμεσα στην εφαρμογή των κανόνων που προβλέπει ο καονισμός και στις επιπτώσεις στην οικονομική θέση των δικαιοδόχων. Η απάντηση είναι όχι. Παραδείγματα. Είναι η ρήτρα μία ανταγωνισμού ε, η απαγόρευση της πολλαπλής δικαιοχρησίας και όλες οι υποχρεώσεις αγοράς ε, που βαραίνουν τους δικαιοδόχους. Παραδείγματο χάρη η απαγόρευση για την πολλαπλή δικαιοχρησία. Υπάρχει αναλογικότητα τη στιγμή που ο δικαιοπάροχος αφού αρνήθηκε να συνεργαστεί ή μάλλον να συνεργαστεί με τον δικαιοδόχο σε περίπτωση που ανοίξει δεύτερο και τρίτο μαγαζί αυτός μπορεί να ανοίξει δεύτερο ή τρίτο μαγαζί, ενώ ο δικαιολόγος δεν μπορεί και αυτό το υποστηρίζει ο κανονισμός. Δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα λοιπόν. Όπως είπε και η υπόθεση προνάψια, ο κανονισμός λέει ότι περιοριστικές ρήτρε σε συμφωνίες δικαιοχρησίας δεν παραβιάζουν του, τους κανόνες του ανταγωνισμού στο βαθμό που χρειάζονται για τον δικαιοπάρχο προκειμένου να προστατεύσει την τεχνογνωσία του, την ταυτότητά του και τη φήμη του δικτύου του. Αυτοί οι περιορισμοί όμως μπορεί να μην πάνε, ε, μπορεί να πηγαίνουν πέρα από το απολύτως απαραίτητο. Έτσι. Οι κατευθυντήριες ε, γραμμές θεωρούνται όμως ότι ε, επιβάλλουν πολύ βαριές υποχρεώσεις για να προστατεύσουν τα, τα συμφέροντα του δικαιοπαρόχου. Δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση είναι υπέρ του δικαιοδόχου. Δεν υπάρχει πουθενά αναλογικότητα με πολύ λίγες εξαιρέσεις, ειδικά με την περάτωση της συμφωνίας. Ο δικαιοδόχος ε, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει ότι η τεχνογνωσία του δικαιοπαρόχου δικαιολογεί το να κλείσει αυτό στην επιχείρησή του. Στο βαθμό που δεν ε, επιθυμεί να συνεχίσει τη σχέση με τον δικαιοπάρχο μετά το τέλος, ας πούμε, της ε, σύμβασης. Έχω παραδείγματα από τους Βέλγους συναδέλφους μερικοί ε, δικαιοδόχοι να αλλάξουν τη φόρμουλα μετά το τέλος του, την περάτωση του συμβολέου του, ε, γιατί έχει, κάνει, έχει περάσει συγχώνευση με τον δικαιοπάρχο. Αυτό όμως δεν το επιτρέπει το δίκαιο ανταγωνισμού. Τη στιγμή που και ο Πάρχος αποφασίζει να αλλάξει τη φόρμουλα του, θα πρέπει να σταματήσει για μία περίοδο ενός έτους. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι λόγος για να παραβιάσει κανείς τα συμφέροντα του δικαιοδόχου. Ο δικαιοδόχος υποτίθεται ότι είναι ελεύθερος να πάει στο δικαστήριο. Αλλά αυτό αγνοεί τις δυσκολίες που έχουν, τις πρακτικές δυσκολίες οι δικαιοδόχοι. Ε, μερικές φορές δεν υπάρχει νομοθεσία που θα τους προστατεύσει και καθίσταται εντελώς αδύναμος ο δικαιοδόχος. Και μην ξεχνάτε βεβαίως και το κόστος να πάει στο δικαστήριο. Ε, και ο, υπάρχει και το στοιχείο του φόβου. Η απλή λύση είναι να απαγορεύσουμε πάντα τη ρήτρα της μης, του μη ανταγωνισμού μετά το πέρας της σύμβασης, εκτός και αν ο δικαιοπάροχος αποδείξει ότι υπάρχει παραβίαση της τεχνογνωσίας του. Και δεν θα πρέπει να περιμένουμε το 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού. Αυτό μπορεί να επιληθεί με άμεση προσαρμογή ε, των ε, κατευθυντήριων γραμμών στις ανάγκες. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Επίσης, η... το Κοινοβούλιο το 2013 ζήτησε να γίνει μια αναθεώρηση με ένα χαμηλό κατόφλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει μεταξύ άλλων πραγμάτων να ξανασκεφτεί τις ε, υπάρχουσες εξαιρέσεις από το δίκαιο ανταγωνισμού για τα συμβαλόμενα μέρη που έχουν μερίδιο της αγοράς λιγότερο από το 30%. Δυστυχώ όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, επίσης, θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στα συμπράσματα της μελέτης, ότι οι ειδικέ κατευθυντήριες γραμμές για τη δικαιοχρησία, για, την άμεση, ε, για τον άμεσο ανταγωνισμό ε, του δικαιοδόχου έναντι του δικαιοπάροχου λείπουν. Επίσης, ε, την ψηφιοποίηση, την αγνοεί εντελώ ο κανονισμό, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οδηγεί σε ανταγωνισμό ανάμεσα στον δικαιοδόχο και στον δικαιοπάροχο, ειδικά εάν αφορά τον τομέα της αγοράς του δικαιοδόχου. Η διαφάνεια σε σχέση ε, με τη διανομή και την κατανομή των κερδών λείπουν. Και έχουμε παρατηρήσει ότι και οι μεν και οι δε ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο και ο δικαιοπάροχος στον δικαιοδόχο και αντίστροφα. Ε, επίσης, ε, στοιχεία των καταναλωτών. Δεν είναι σαφέ ποιο μπορεί, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των καταναλωτών και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που ε, λαμβάνει ας πούμε ο δικαιοδόχο, Ο δικαιοπάροχο ε, εκπεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα ε, και χρησιμοποιεί τα δεδομένα ε, που, έχουν συλλεχθεί για να προσεγγίσει του πελάτε. Ακόμα και πελάτε που ήταν αρχικά κυρίω πελάτε του δικαιοδόχου και δεν το ξέρει καν ο δικαιοδόχο μερικές φορές. Σε μια τέτοια σχέση οι δικαιοδόχοι θέλουν να συμμετάσχουν, να συλλέξουν τα στοιχεία λοιπά, υπό τον όρο ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να υποφεληθούν και αυτοί από τα στοιχεία. Και να υποφεληθούν και από τις πληροφορίες που απορρέουν από τα δεδομένα αυτά. Επομένως, ο κανονισμός για τα ψηφιακά στοιχεία ε, θα πρέπει να ο κανονισμό θα πρέπει να επεκταθεί και στα ψηφιακά στοιχεία τη σχέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει μια καλή συνεργασία ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και στη Γενική Διεύθυνση ε, Grow. Παρότι ε, οι υπηρεσίε και στι δύο γενικέ διευθύνσει είναι πολύ συνεργάσιμε και η ΜΕΝ και η δε λένε ότι κοιτάξτε η άλλη υπηρεσία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ε, έχουμε από τη μία τον ανταγωνισμό και από την άλλη κατάχρηση τη ισότιμης των ισότιμων όρων, να πούμε. Ο, η Επίτροπος ε, απάντησε θετικά στο, στην πρόσκλησή σας να προωθηθεί η συζήτηση για τα θέματα της δικαιοχρησίας. Θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Ε, είναι η αυτορύθμιση η λύση. Εγώ είμαι συντάκτης, ε, μία από τους συντάκτες του Ολλανδικού κώδικα και τον υποστηρίζω. Είναι σαφώς ότι ο NFC, ο κώδικας αυτός, είναι συμβασμός μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Με την εισαγωγή του κώδικα έχουμε ε, ένα πιο υγιές και πιο ισορροπημένο περιβάλλον στον τομέα της δικαιοχρησίας. Ε, ικανοποιεί αυτός ο, κώδικας. Αλλά η εισαγωγή νομοθεσίας που υποχρεώνει το να εφαρμόσουμε τον κώδικα είναι ο επόμενος σκοπός μας, δεδομένου του ότι οι, οργανώσεις, οι Ολλανδικές Οργανώσεις ε, Δικαιοπαρόχων αποφάσισαν να μην δεχτούν τον κώδικα, παρότι το ζήτησαν οι οργανώσεις των δικαιοδόχων. Ε, επομένως, χρειαζόμαστε νομοθετική υποστήριξη. Και αυτό το αποδεικνύει και η μελέτη, την ανάγκη αυτή. Ε, εθελοντική κωδική B2B μεταξύ επιχειρήσεων. Θα είναι καλό τρόπο για να αντιμετωπιστούν οι εντάσει όταν υπάρχουν αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Αλλά παν, μετά από πάνω από 40 χρόνια στη δουλειά, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικαιοχρησίας στην πραγματικότητα δεν υιοθετήθηκε υποχρεωτικά ούτε από τα δικαστήρια, ούτε από το τομέα της δικαιοχρησίας, τον κλάδο δηλαδή, ούτε από τις τράπεζες. Και δεν έχει συνεισφέρει ε, στο να κατευνάσει τις εντάσεις στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Δικαιοχρησίας δεν εκπροσωπεί τους δικαιοδόχους επίσης. Ήθελα να το πω αυτό. Κοιτάξαμε όλες τις οργανώσεις και τις ιστοσελίδες τους και με ενδιαφέρον είδαμε ότι μόνο μια τέτοια οργάνωση, η Βρετανική, εκπροσωπείται, ακόμα μία εξαίρεση των Βρυτανών. Υπάρχουν και άλλες δύο εξαιρέσεις στη Σουηδία. Οι δικαιοδόχοι αυτόματα είναι μέλη και στη Δανία υπάρχει δυνατότητα ε, οι δικαιοδόχοι να γίνουν μέλη, αλλά δεν έχουν δικαιώματα ψήφου στις οργανώσεις των δικαιοπαρόχων. Επανέρχομαι στον ε, Ευρωπαϊκό Κώδικα Δικαιοχρησίας του 2016. Είναι μονόπαντο που το έχουν καθορίσει οι δικαιοπάροχοι χωρίς να έρθουν σε επαφή με τους ε, εταίρους τους, με τους δικαιοδόχους δηλαδή, με τους ομολόγους τους. Εάν ενδιαφέρεστε για τα σχόλιά μας για το νέο κώδικα, με μεγάλη χαρά σας τα δώσουμε. Να αναφέρω τελειώντας ότι η λέξη ο, υποχρεώσεις των δικαιοπαρόχων στον παλιό κώδικα αναφέρονται στο νέο κώδικα ως δεσμεύσεις. Και η συμφωνία που έλεγε το 5-2 ότι ε, η συμφωνία και η υπογραφή τους θα πρέπει να... ή μάλλον η μαλλον θα πρέπει να γράφεται γραπτός, αυτό δεν υπάρχει πια στο νέο κώδικα. Είναι αθέμητη πρακτική το γεγονός ότι δεν έχουμε γραπτός αυτές τις δεσμεύσεις. Η επόμενη διαφάνεια. Η αυτορύθμιση ε, είναι λύση μόνο αν συνοδεύεται από υποχρεώσεις. Νομική προστασία της θέσης των δικαιοδόχων σε, στην προσυμβατική και στη συμβατική φάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και υποστηρίζω αυτά τα συμπεράσματα, τα σχετικά συμπεράσματα της μελέτης. Όπως ε, δείχνει και η διαφάνεια, μπορείτε να βρείτε κάποια από τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σε ένα κανονισμό και η ανάγκη ε, του να μπαίνουν κάποια πράγματα γραπτός, αυτό είναι εκ των όνου κάνευ. Επίσης, ε, το δίκαιο ανταγωνισμού ή το ιδιωτικό δίκαιο. Επανέρχομαι στην μελέτη. Ε, υποστηρίζουμε το συμπέρασμα ότι τα μέτρα του δικαίου του ανταγωνισμού θα πρέπει να αξιολογηθούν όχι μόνο από τη σκοπιά της αγοράς και της ολοκλήρωσης, αλλά και από τη σκοπιά των σχέσεων που υπάρχει. Μία δικαιοχρησία δεν είναι μια σύμβαση ανάμεσα, μια σύμβαση δικαιοχρησίας δεν είναι μια συμβαση αναμεσα μια συμβαση δικαιοχρησια ανάμεσα σε δύο ισότιμα μέρη. Θέλω να πω και κάτι θετικό τελειώνοντα όμω. Θέλω να σα πω ότι ένα ισορροπημένο κανονισμό για την ε, δικαιοχρησία είναι καλό για του επιχειρηματίε, για του καταναλωτέ, για του τοπικού προμηθευτέ, για την καινοτομία, για την απασχόληση. Επομένω, α μην χάνουμε χρόνο και α αρχίσουμε τώρα να ρυθμίσουμε σωστά τα πράγματα με σωστούς κανονισμούς. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού περάσουμε στον επόμενο εμιλητή, έχω ένα διαδικαστικό και για τους Γερμηνείς. Επισήμως πρέπει να τελειώσουμε στις 5.30. Επειδή καθυστερούμε, δεν θα έχουμε διερμηνία πλέον μετά τις 5.30. Πρέπει να αφήσουμε την αίθουσα. Εάν λοιπόν θέλετε να συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε μετά τις 5.30 αλλά χωρίς διερμηνία. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε και τους ε, δικαιοδόχους που βρίσκονται στην αίθουσα για να μας πούν τη δική τους ιστορία. Μιας και μιλάμε για δυτικό δίκαιο. Ο επόμενο εμπειρογνώμων είναι ο κύριος Οντάβια, η κυρία Οντάβια Μπερναντία, δόκτωρ Οντάβια Μπερναντία. η οποία είναι ε, ειδική στη σχετική εταιρεία και μέλος της ομάδας για τον Ευρωπαϊκό Εμπορικό Κώδικα και τις σχετικές συμβάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ εκπροσωπώ τη δική μου εταιρεία. Διότι εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο του Σαν Σεμπάν, αλλά είμαι και νομικός στην Ισπανία και η προγνωμοσύνη μου προέρχεται από τη συμμετοχή μου στην εταιρεία αυτή και κυρίως ε, στην ομάδα εργασίας για τον αστικό κώδικα και την ομάδα Άμστερνταμ το 2006. Υποβάλαμε τις αρχές μας για την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμβάσει διανομή και την δικαιοχρησία. Οι λύσει υπάρχουν γιατί τι προτείναμε ήδη το 2006. Όμω, ήταν οι βασικές αρχέ που να διέπουν τις ε, συμβάσει δικαιοχρησία. Στην εταιρεία μου έχω κάποια εμπειρία, ιδίω με του δικαιοδόχου. Και μια και εδώ πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο απλά, ε, μερικέ από τι δικέ μου εμπειρίε είναι ότι όταν πηγαίνω στο φούρνο κάθε πρωί θέλω να είναι το ψωμί μου άσπρο. Ε, δεν θέλω ολική αλέσεω. Η Ελένα που είναι η φουρνάρισα μου είπε ότι δεν μπορεί να έχει δημητριακά καθημερινά διότι έχει εταιρεία δικαιοχρησία και πρέπει να αγοράζει αποκλειστικά από την πηγή τη δικαιοχρησία, από το δικαιοπάροχο. Αλλά δεν έχει πάντοτε λευκό ψωμί ο δικαιοπάροχο να τη δώσει και οπότε δεν έχει άλλο τρόπο, δεν έχει επιλογή παρά να πει στον καταναλωτή σήμερα δεν έχει λευκό ψωμί. Λυπούμε. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξω φούρνο. Μετά έχω μια φίλη που άνοιξε εταιρεία δικαιοχρησία για, για μια σχολή μουσική. τελευταία φορά που πήγαμε από τι γίνεται, διαφήμιζε υλικό από το 2014. Ρώτησα γιατί δεν έχει πιο πρόσφατο υλικό. Είπε γιατί έχω αποκλειστική υποχρέωση να περνάω το υλικό από τον δικαιοπαροχό μου. Όμω δεν μου δίνει πιο επικαιροποιημένο υλικό. Δεν μπορώ να πάρω παλού. Next, ε, συγγνώμη, δίπλα στο σπίτι μου υπήρχε ένα σούπερ μάρκετ, ένα ντία. Εδώ είχαν την υποχρέωση να αγοράζουν μόνο από την πηγή των δικαιοπαραχών, λόγω χάρη προϊόντα στα 80 λεπτά, τα προϊόντα αυτά για ένα ευρώ τα αγόραζαν και πληρώναν το δικαιοπάροχο εκ των υστέρων, κάνοντα και την προώθηση και τη διαφήμιση αυτών των προϊόντων με 60 λεπτά. Ο ιδιοκτήτη του Ντία δίπλα στο σπίτι μου πτώχευσε βέβαια. Και είναι ένας από τους 80 δικαιοδόχους που έχει προσφύγει στα ισπανικά δικαστήρια κατά του δικαιοπαρόχου του. Το ίδιο 30 ε, άλλοι εμπορευόμενοι στην Γαλλία και την Πορτογαλία. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί είμαστε όλοι θετικοί ω προ την δικαιοχρησία. Αλλά βλέπουμε να υπάρχουν και προβλήματα. Υπάρχουν τριγμοί στι σχέσει δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Δεν έχουν αρκετή δύναμη διαπραγμάτευση. Είναι συνήθω οι πιο ισχυροί δικαιοπάροχοι γιατί έχουν τη φόρμουλα τη δικαιοχρησία στα χέρια του και αυτό είναι σαφέ και πρέπει να γίνεται σεβαστό. Όμω πρέπει να επιβληθούν ε, περιορισμοί και στους δικαιοδόχους. Δεν μπορούν να τους ε, υποβάλλουν απλείς, ε, μάλλον μπορούν να υποβάλλουν στην ελευθερία τους κάποιες κάποιους περιορισμούς, αλλά όταν αυτή η, αρμοδιο, η εξουσία χρησιμοποιείται μάλλον υπερβολικά τα καταχρηστικά ει βάρο του δικαιοδόχου υπάρχει πρόβλημα. Πάω στη σελίδα 12 γιατί τα πάντα έχουν ε, υποθεί ήδη και θα επικεντρωθώ στι πολιτικέ επιλογέ. Τι μπορεί να κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα δράση. Γνωρίζουμε και η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εγκεφουστών ξέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα. Και υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε απευθεία στου δικαιοδόχου και στι μικρομεσαίε κυρίω είτε είναι μικρομεσαίες είτε μικρομεσαίες που συνεργάζονται με άλλες μικρομεσαίες. Τότε οι δικαιοδόχοι πρέπει να έχουν την απαραίτητη, τις απαραίτητες πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για να μπορούν να οργανώσουν την επιχείρησή τους. Πάντοτε υπάρχει έλλειψη ισορροπία βέβαια. Ε, σε περίπτωση μεγάλου δικαιοπαρόχου, παρόλο που δεν είναι αυτό το σύνηθε, θα έλεγα ότι είναι μειονότητα. Πολλέ φορέ φοβούνται ε, οι δικαιοδόχοι να προσφύγουν κατά του δικαιοπαρόχου, διότι θα πτωχεύσουν, η διάρκεια της δραστηριότητα τους εξαρτάται ε, από την ε, καθημερινότητα της προσφοράς υπηρεσιών, δεν μιλάμε τώρα για τους μεγάλους δικαιοδόχους, ε, δεν έχουν αρκετέ επιλογές που έχουν δικαιοπάροχοι. Ως προς την υποεκπροσώπηση των δικαιοδόχων, η Ομοσπονδία των Δικαιοπαρόχων, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αλλά είναι ότι είναι φωνή του κλάδου. Ακόμη και όταν είπε η Μάρτα προηγουμένω, δεν είναι σύμβαση η αμφίπλογη. Διότι είναι δίκτυο η σύμβαση, είναι δικτυακή. Ένα ο δικαιοπάροχο και πολλοί δικαιοδόχοι που συνδέονται μαζί του. Οπότε πρέπει να ακούγεται τη φωνή και των δύο πλευρών, να γνωρίζουν ε, τα προβλήματα και να μπορούν και να τα επισημάνουν. Μια άλλη παρατήρηση, το διασυνοριακό στοιχείο στη δικαιοχρησία. Αυτό δεν το είδα στη μελέτη τη ΣΥΜΚΟ και νομίζω ότι είναι μείζον ζήτημα. Η δικαιοχρησία σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα δίκτυο όπου διάφορα κράτη από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης μπορούν να διασυνδεθούν η διατήρηση της φήμης του δικτύου, της καλής φήμης, απαιτεί ομοιομορφία στη λειτουργία του. Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο διασυνοριακό. Ίσως να μην με ακούγατε από την αρχή της συνεδρίασης. Πείτε με αν δεν με ακούτε. Πού ήμουν. Το διασυνοριακό στοιχείο στις σχέσεις δικαιοχρησίας. Ο δικαιοπάροχος έχει πολλούς δικαιοδόχους. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε μόνο χώρο δικαιοχρησία, αλλά να πάμε παραπέρα και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σε όλα τα κράτη-μέλη, τέλος πάντων σε πολλά. Υπό αυτήν την έννοια πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στην παροχή των υπηρεσιών. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονό ότι οι σε πολλά κράτη-μέλη σε διαφορετικά κατημέλη θα πρέπει να την χάνουν ίσε μεταχείριση και ίδιε μεταχείριση. Γι' αυτό είναι σημαντική η ομοιομορφία στο δίκτυο. Αυτέ οι δυσκολίε μπορεί να έχουν επιπτώσει στην εσωτερική αγορά ή και στην ε, ευημερία του καταναλωτή. Δηλαδή, σκεφτείτε το λευκό ψωμί που θέλω να αγοράζω που δεν μπορώ να το βρω γιατί δεν το παρέχει ο δικαιοπάροχο. Επίσης ε, για τον ε, δικαιοπάροχο. Αυτά που συμβαίνουν τώρα τουλάχιστον στην Ισπανία, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλα συστήματα. Αλλά η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δικαιοδόχοι, οι πρώην δικαιοδόχοι, που θεωρούν ότι έπεσαν αντικείμενο εκμετάλλευση ή ότι πτώχευσαν και ότι είναι θύματα, ε, με πολύ μεγάλες συνθήκες στρες πρέπει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και μετά πολλές φορές επιλέγουν να υποβάλουν συλλογικές προσφυγές σε συνεργασία με άλλους δικαιοδόχους, οι οποίοι θα πλήξουν το δίκτυο του δικαιοπαρόχου. Μην ξεχνάμε, αν πάει κανείς στο ίντερνετ και κοιτάξει για τέτοιες αξιώσεις δικαιοχρησίας, είναι πάρα πολλές ε, οι περιπτώσεις ανθρώπων που πτώχευσαν και ε, δυσφημούν το δίκτυο του δικαιοπαρόχου του δικαιοπαρόχου, έχουν στραφεί εναντίον του, το οποίο μπορεί να έχει πολύ κακές συνέπειες για τη φήμη του δικαιοπαρόχου. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιος είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιτρέψουμε στη φωνή των δικαιοδόχων να ακουστεί. Δεν ακούγονται αρκετά όπως πάνε περισσότεροι. Πρέπει να ενισχυθούν οι ενώσεις τους με ενώσεις όπως η Γάμη, που είναι μία ένωση και άλλες. Οι αξιώσεις εμπιστευτικότητας είναι σημαντικές για τη δικαιοχρησία. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε τις πληροφορίε που χρειαζόμαστε χωρίς να ε, υποκύπτουμε στις απαιτήσει άρσης ή όχι το πολίτη. Επίσης, μπορούμε να βοηθήσουμε ε, εάν ε, καθησυχάσουμε τους φόβους των ε, δικαιοπαρόχων του κλάδου. Λόγω χάρη, εκφράζοντας την ιδέα ότι αν συνεχίσουν έτσι με τις δικαιοχρησίες, θα καταλήξουμε σε περισσότερες συλλογικέ προσφυγές και αμάβρωση της φήμης του δικαιοπαρόχου στο ίντερνετ. Για τους ισότιμους κανόνες, εφόσον αυτό ισχύσει, μπορούμε να ρωτήσουμε τους ενδιαφερομένους τι άποψη έχουν και οι ίδιοι. Ε, η συλλογή πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Ε, υπάρχουν ήδη πολλέ, διότι αθέμετε πρακτικέ για την επιστημιστική και μία λυσίδα μα δείχνει πώ λειτουργεί η δικαιοθεσία. Και μετά υπάρχουν άλλε αθέμετε εμπορικέ πρακτικέ, UTPs, οι οποίε προσυδειάζουν στον τομέα τη δικαιοθεσία. Στο έγγραφο κιόλα ενδιαφέρονται αναφέρονται διαφορετικέ πολιτικέ επιλογέ που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Λόγω χάρη να ρωτήσουμε του ενδιαφερομένου ποια κατεύθυνση θέλετε εσεί να ακολουθήσουμε. Η μία είναι μηδέν παρέμβαση. Αυτό μπορεί να απαντήσουν αν βρίσκονται σε ίσε περίπου θέσει. Δεν υπάρχει λόγο παρέμβαση. Έχουν περίπου τέτοια συμφέροντα. Εγώ θα πω αυτό που μόλι είπα. Ότι αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα. Για του δικαιοδόχου αλλά και για πολλού δικαιοπαρόχου. Επίσης, θα μπορούσαμε να βρούμε μια ε, ενδιάμεση λύση. Επαναπροσαρμογής. Αξιοποίηση των των κανονισμών. Και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον ανταγωνισμό πρέπει να ξαναπάμε στην απόφαση προνούψια, διότι επιτράπηκαν εξαιρέσει που ήταν καθοριστική σημασία, περιορισμοί που δεν θα προστατεύσουν απλώ τη φόρμουλα. Οι υποχρεώσει υποχρεωτική αγορά. που όμως δεν είναι οι ίδιες ως προς τις υποχρέωσεις προμήθεια του δικαιοπαραγωγού, οπότε υπάρχει πρόβλημα στρεβλής λειτουργίας του δικαίου ανταγωνισμού. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό. Η αυτορύθμιση επίσης είναι σημαντική. Και θα μπορούσαμε να αποφεληθούμε για το Ευρωπαϊκό Κώδικα, ο κώδικα τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Δικαιοκρισία είναι πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ ε, αξιόπιστο για το πώ μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μα. Απλώς το πρόβλημα που βλέπουμε αυτόν τον κώδικα είναι ότι δεν εκπροσωπούνται αρκετά οι δικαιοδόχοι και είναι απλώς ένα στοιχείο ε, βιτρίνας, δηλαδή χρησιμοποιείται μόνο όταν περάσουν στην Ένωση των Μελών και οι δικαιοπάροχοι. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί ε, επιβολής του εφαρμογή του. Οπότε έτσι κι αλλιώ χάνουμε το στόχο. Πρέπει να υπάρξει ένα εξισορροπημένο σύστημα ώστε οι δικαιοδόχοι να συμμετάσχουν στου στους φορείς αλλά όπως είπε και η κυρία Τσόπρα, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Ε, έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και ευθύνε. Είναι πρόβλημα του συστήματο αυτό όμω. Θέλουμε δικαιοπαράχου και δικαιοδόχου που πρέπει να συνομιλήσουν, να έρθουν και να ανοίξουν το στόμα του. Μια άλλη λύση Όπως λέει και η μελέτη της ΣΥΜΚΟ, από τις υπάρχουσες οδηγίες πρέπει να δούμε τι ισχύει για τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές. Να διπλασιάσουμε τις υποχρεώσεις και να τις ενισχύσουμε. Τελευταία πολύ επιλογή λίγο ακραία. Εκ του μηδενός, να ε, θεσπίσουμε νέες αρχές για την σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυνατόν. Νομίζω επόμενη, η επόμενη διαφάνεια θα το ξεκαθαρίσει. Επόμενη. Πρέπει να πάτε στην διαφάνεια περιθμών μισό λεπτό, 19. Η δυνατότητα να υπάρξουν αρχές ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή εφόσον μπορούμε να βασιστούμε σε κάποια μοντέλα με το κώδικα συμπεριφοράς, με αυτά που προέκυψαν από την Ολλανδία, τον ε, κώδικα του Υπουργείου για τη Δικαιοχρησία. Μετά από τόσους γύρους συζητήσεων, καλό θα ήταν να ακούσουμε τουλάχιστον την άποψη των δικαιοδόχων και να ξαναδούμε τις αρχές του εμπορικού δικαίου των, ε, ε, και τις αρχές που μπορούν να διέπουν τις συμβάσεις διανομή. Και αυτές οι αρχές βασίζονται σε αποκρίσεις κάτι κράτη-μέλη και την νομολογία και δίνουν τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια σταθερή βάση με γενικές αρχές και ειδικότερε για το πώς οι δικαιοπάροχοι και οι δικαιοδόχοι θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση πρόκειται για μια πρόταση που θα πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενδεχόμενη πρόταση θα μπορούσε να είναι, όπως τη βλέπω εγώ, για ευρωπαϊκές αρχές, ο ορισμός της δικαιοχρησίας, κάτι που ε, εμφανίζεται στον κανονισμό. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη δικαιοχρησία, αλλά πρέπει να κάνουμε τι απαραίτητε διακρίσει. Ποια είναι η βιομηχανική δικαιοχρησία, ποια είναι αυτή των υπηρεσιών, ποια είναι η εμπορική. Για ποια μιλάμε. Και μετά πρέπει να βρούμε γενικέ αρχέ. πιο συγκεκριμένε για την εξισορρόπηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Και ένα μηχανισμό ένδικων μέσων που να επιτρέπει την διάρκεια και παροχή. Όλα αυτά για να πω ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε και τη γνώμη του κόσμου, να ακουστεί η φωνή τους, διότι με βάση αυτές τις αρχές μπορούν να μας πούν ποιες φόρμουλες τους φαίνονται πιο αποτελεσματικέ. το αν θα υπάρξει αυτορύθμιση ή λύση ιδιωτικού δικαίου και τέλο πάντων ήδη συμπεράσματο να πω ότι η μελέτη ΙΜΚΟ προσφέρει και έχει εντοπίσει τα βασικά προβλήματα στην, στα δίκτυα ειδικοχρησία. και τρόπους ε, ε, να προχωρήσουμε στο όλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Όσο περισσότερο ακούω, τόσο περίπλοκο, τόσο πιο περίπλοκο γίνεται το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα ήταν εύκολο τελικά να συντάξουμε την έκθεση το καλοκαίρι. Μιλήσαμε λοιπόν για τους δικαιοπαρόχους, για τους δικαιοδόχους, έχουμε επιχειρηματίες ε, στην αίθουσα, οπότε θα δώσουμε προτεραιότητα σε όσους ε, ε, κατέχουν εταιρεία, όσους είναι δικαιοδόχοι. Εμείς είμαστε δικαιοπάροχοι η ΕΦΕΦ e μου ζήτησε να δώσω πρώτο το λόγο σε αυτούς που διαχειρίζονται τις εταιρείες ως δικαιοπάροχοι ή ως δικαιοδόχοι για να δούμε τις εμπειρίες σας. Yes, um, good afternoon. Καλησπέρα σας. Michael Air ε, επιχειρηματίας δικαιοπάροχος με βάση τον Ηνωμένο Βασίλειο και είμαι πρόεδρος της, ε, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Δικαιοπαρόχων και είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής ε, ε Ομοσπονδίας Δικαιοχρησίας και αν υπάρχουν ερωτήσεις ευχαρίστω να σας απαντήσω. You, you any but... Δέχεστε ερωτήσεις. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε την εμπειρία των επιχειρηματιών, την ε, πρακτική τους εμπειρία, είτε ως δικαιοπάροχοι είτε ως δικαιοδόχοι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα σας ρωτήσουμε εμείς, ε, θα σας θέσουμε εμείς ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Νταγιόν που μου δίνετε την ευκαιρία. Νομίζω το είπατε στην αρχή ότι αυτή είναι μια ε, πολύπλοκη έκθεση. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι αρκετά μακροσκελής και επίσης δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ε, ότι ταυτόχρονα ε, αυτή η έκθεση ε, από αυτή την έκθεση λείπουν πολλά στοιχεία. Έχουμε τις συζητήσεις για το Brexit, για το Remain και εδώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολλές εκθέσεις λοιπόν με πολλά στοιχεία με πολύ ίσως άσχημα αποτελέσματα. αποτελέσματα. Εγώ θα, θα ήθελα να προτείνω σε όλους την έκθεση της, για την έλλειψη της, της διαφάνειας στην αγορά, που ουσιαστικά λέει ότι δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Ε, νομίζω λοιπόν ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά την έρευνα, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Και βεβαίως εγώ πιστεύω ότι στη δική σας την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας θα πρέπει αυτό να το καταγράψετε. Ναι, η Ανέτα θέλει το λόγο. Ναι, ναι, ναι, επανέλθω παρακαλώ αν μπορώ. Yes, thank you, uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εμένα με προειδοποίησαν ότι αν πω ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα μπαίνω σε πολύ επικίνδυνα ύδατα. Ε, χρειάζεται όμως να γίνει περισσότερη έρευνα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι η έκθεση δεν περιλαμβάνει τα ε, επαρκή στοιχεία όπως υπόθηκε. Αυτό που μου ε, κάνει εντύπωση μετά από τόσες ώρες συζήτησης και βεβαίω, εντάξει, μπορείτε να, ε, μπορεί να μην σα αρέσει αυτή η προσέγγιση τη συζήτηση με του ανθρώπου, αλλά αν δεν υπάρχουν άλλα, άλλη βάση για την σύνταξη τη έκθεση, είναι η μόνη διαλλακτική που έχουμε. Μετά από μήνε, λοιπόν, ε, που δουλέψαμε πάνω στο το φάκελο για τη δικαιοχρησία, εγώ είμαι σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών της Ολλανδίας και η δική μας εμπειρία ήταν ε, σημαντικά σχεδόν πανομοιότυπη. Οπότε με ενθαρρύνει η συζήτηση που κάναμε με την εκπρόσωπο του ε, Ολλανδικού Υπουργείου Οικονομικών, για να πω αυτά που λέω. Και επειδή δεν έχω απτά αποτελέσματα, ε, δεν έχω πρόσβαση εγώ σε τέτοιου είδου συμβάσεις, και το είπα σαφώς, παρόλα αυτά, ομοιότητες υπάρχουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Να επανέλθουμε σε εσά. Ναι, ευχαριστώ. Στην αρχή της παρουσίασής σας μας παρουσιάσατε έναν κατάλογο με τις χώρες που πήρατε πληροφορίες, από τις οποίες πήρατε πληροφορίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν στον κατάλογο αυτό. Με εκπλήσει πραγματικά που δεν βρήκατε τέτοιε συμβάσει δικαιοχρησία. Είπατε ότι είχατε πολύ μεγάλο πρόβλημα να, να, ε, βρείτε τέτοια στοιχεία. Έχουμε 150 δικαιοπαρόχου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με ευχαρίστηση θα σα έδιναν τι συμβάσει του. Αν πάτε μάλιστα στην ιστοσελίδα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μα σε PDF οι συμβάσει αυτέ. από ό,τι ακούσαμε και σήμερα το απόγευμα, υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία ε, δικαιοδόχων που είναι ε, δυσαρεστημένοι. Εμείς κάναμε μια ανεξάρτητη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, το 97% των δικαιοδόχων ήταν αρκετά ικανοποιημένοι με τη συμβατική σχέση που έχουν με τους δικαιοπαρόχους. Οπότε αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει τουλάχιστον στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και η, η εμπειρία μου από το EFF δεν είναι καθόλου όμοια με αυτή της, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ίσως μια προκατάληψη προς κάποια πολύ μικρή μερίδα εκπροσώπων της μιας της άλλης πλευράς. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι έχει, έχει διαραγεί η σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Yes, thank you very much for... Ευχαριστώ. Να σας διευκρινίσω το εξής εδώ. Το πεδίο της έρευνας με τις εννέα χώρες που σας παρουσίασα και που ερευνήσαμε, ε, αυτό το πεδίο το καθόρισε το Κοινοβούλιο. Εμείς δεν είχαμε λόγο στην επιλογή των χωρών. Ε, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του Κοινοβουλίου. Μάλιστα ξέχασα και το επίσημο όνομα του κειμένου που λάβαμε. Ακολουθήσαμε τους όρους αναφοράς. Του όρους αναφοράς με βάση οποίου μα ανατέθηκε η μελέτη. Κρίμα είναι. Αν πάντως συνεχιστεί αυτή η έρευνα, ε, σας λέμε από τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν ε, πρόθυμο να συνεργαστεί. Σίγουρα θα κοιτάξουμε πάντως την ιστοσελίδα σας πριν γράψουμε την έκθεση. Ο επόμενος ομιλητής. Είμαι σαν ανεξάρτητος λιανέμπορος στην Ολλανδία Είμαι ε, δικαιοδόχος εδώ και 28 χρόνια. Λατρεύω τη δικαιοχρησία, είναι καλό σύστημα, μπορείς να συνεργαστείς, μπορεί να είναι εποφελές και για σένα και για τον ομόλογό σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να υπάρχει και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δικαιοδόχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και από αυτά που άκουσα σήμερα, Ορισμένοι αγνοούν αυτά τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα των δικαιοδόχων. Είναι αδύνατο σε ένα σύστημα. Αν, α πούμε, είσαι δικαιοδόχο και είσαι ένα μαγαζί. Ο δικαιοπάροχό σου να περιφέρεται, ας πούμε, με ένα φορτηγό και να πουλάει ε, τα ίδια προϊόντα τα οποία είσαι εσύ στο μαγαζί σου και να παραδίδει τα προϊόντα στους δικούς σου πελάτες στην περιοχή σου. Έχεις κάνει συμφωνία με αυτόν τον άνθρωπο ότι μια συγκεκριμένη περιοχή είναι δική σου, δική σου ως δικαιοδόχου. Αυτό λένε, το λένε και οι συμβάσεις που υπογράφεις. Είναι πολύ παράδοξο που ο δικαιοπάροχος οδηγεί, ας πούμε, με ένα φορτηγό στη δική σου περιοχή και με αυτόν τον τρόπο χάνεις. Δεν κάνεις πωλήσει, χάνεις κέρδη δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο και σε περίπτωση που γίνεται δεν είναι δίκαιο. Επίσης δεν είναι δίκαιο όμως όταν ένα δικαιοδόχος πτωχεύει, ένας νέος δικαιοδόχος να μπορεί να αγοράσει σε ψηλές τιμές τα αγαθά και το μαγαζί και όλο τον εξοπλισμό. Τα ψυγεία, πληρώνοντας πολλά λεφτά και μετά από λίγα χρόνια ή λίγου μήνε να πτωχεύει και αυτό. Δηλαδή να, έχουμε τη μία πτώχευση μετά την άλλη των δικαιοδόχων. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ. Είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα. Δεν μου αρέσει η δικαιοχρησία. Εδώ μιλάμε για δικαιοδόχου που θέλουν να είναι σίγουροι ότι αυτό το πράγμα θα γίνεται συνέχεια. Δηλαδή θα το ένα με τον άλλον, α πούμε. Και υπάρχει και συμφωνία ανάμεσα στους δύο για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Το θέμα δεν είναι αν είναι καλή ή κακή η δικαιοπάροχη. Το θέμα είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, να δούμε πού είναι τα προβλήματα και να εξασφαλίσουμε ότι όπως και στην Ολλανδία που έχουμε τον Ολλανδικό κώδικα, τον NFC, θα βάζουμε στο χαρτί ξεκάθαρα τον τρόπο συνεργασίας. Θα το λέει ξεκάθαρα δηλαδή η σύμβαση. Το τονίζω, είναι σημαντικό αυτό. Και ο δικαιοδόχος και ο δικαιοπάροχος να συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Και αν δεν μπορούν να συνεργαστούν, τότε χρειαζόμαστε κάποιο νόμο που θα το επιβάλλει αυτό. Εγώ είμαι ανεξάρτητος επιχειρηματίας, 28 χρόνια και γενικά δεν μου αρέσουν οι νόμοι. Αλλά χρειάζονται και οι νόμοι αν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αλλιώς. Ελεύθερα, αδέσμευτα και χαλαρά. Ευχαριστώ. Στο μεταξύ να ευχαριστήσω και τους. Στο μεταξύ να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς που μας δώσανε λίγο χρόνο παραπάνω. Κανονικά θα πρέπει να περιοριστούμε το, ε, και να σταματήσουμε εδώ τις ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά βλέπω ακόμα έναν να θέλει να θέσει μια ερώτηση. Να τον ακούσουμε και αυτόν. Excuse me. I work for Colroyd, who is one of... Uh, Εργάζομαι για την ε, Colroyd. Conroy, που είναι ε, δικαιοδόχος της ε, στις κάτω Ξεκινήσαμε το 2003 και ανεβήκαμε στις πωλήσει τουλάχιστον 10% για τους δικαιοδόχους και για τη δική μας την επιχείρηση. Τα πάμε δηλαδή πολύ καλά. Θα ήθελα να τονίσω ότι, είχαμε μία, ότι έχουμε μια πτώχευση κάθε χρόνο περίπου και αυτό που έγινε είναι ότι την επιχείρηση την πούλησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, εμείς δεν παρεμβαίνουμε, έχουμε μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να συζητούμε τα διάφορα θέματα. Οι δικαιοδόχοι αποφασίζουν ε, οι ίδιοι αν θέλουν να αγοράσουν. σε μια πλατφόρμα πλειοψηφίας όπου έχουν ε, επιλεγμένους ε, δικαιοδοχούς και αυτό κατά την πείρα μου έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα συνεννόησης μεταξύ δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων. Οι λύσεις που προτείνονται προκύπτουν και αποφασίζονται ε, και προχωρούμε αναλόγως. Έτσι προχωρούμε και ως τώρα δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι πολύ καλή η υγεία της επιχείρησής μας και θέλω να τονίσω ότι Απογοητεύομαι λίγο που βλέπω ότι στον κατάλογο των ανθρώπων με τους οποίους συζητήσατε υπάρχει ο Γλυκαρτής που έχει υποβάλει προσφυγή στο Βέλγιο αλλά χωρίς καμία σπάρ. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό. Πήγαμε να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό, αλλά δεν έχουμε καμία ρήτρα στις συμφωνίες μας ως προς τον ανταγωνισμό και τα σχετικά ζητήματα. Οπότε έλατε να δείτε τι συμφωνίες μας. Υπάρχουν, είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις μελετήσετε. Θα έλεγα να γίνει λίγο πιο ανοιχτό λοιπόν η μελέτη και να μελετήσει ακριβώ τις περιπτώσεις που υπάρχουν και στην αγορά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ε, διαφάνεια την οποία επιδεικνύεται. Υπάρχουν δύο ακόμα, κύριος και κυρία εκεί πίσω. Τελικέ παρεμβάσει. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Τζίλτον Χάρθ, δικαιοδόχο τη κατοχώρε των, σούπερ μάρκετ, κάποιων σούπερ μάρκετ και τριών τροφίμων και έχω μια ερώτηση προς την δόκτωρα Μπενοντίας για τις συμβάσεις. Είπε ότι οι συμβάσεις μπορεί να είναι πρόβλημα ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετές συμβάσεις διαθέσιμες. Εγώ συμμετείχα στη σύνταξη του Ολλανδικού Κώδικα ως δικαιοδόχος και αυτό που παρατηρήσαμε στις συζητήσεις του Κώδικα ήταν ότι το μέγεθος καθορίζεται και μέσω της ε, σύμβασης. και ότι ε, τα ψηλά γράμματα, οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από την κάθε σύμβαση. Πάντοτε υπάρχουν ε, κάποιες ρήτρες ε, μικρές που δεν τις βλέπει κανείς και εφημερούν τον ε, δικαιοπάροχο καταρχήν και είναι δύσκολο να τις αφισβητήσει κανείς σε ομαδικό επίπεδο. Εμείς θεωρούμε πολύ κακό να υπάρχουν καν αυτές οι λεπτομέρειες, οι ρήτρες. Can they also explain how uh, these side letters can be uh, opened for the Πώς μπορούν αυτά να δημοσιοποιούνται στο κοινό ε, και να ε, είναι γνωστές αυτές οι παράπλευρες διατάξεις στα προσθετικά μια σύμβαση. Αυτή είναι η ερώτηση για τους δικαιοπαρόχους και για την ε, δόκτορα Βιβρόφσκα. Πώς βλέπετε το πρόβλημα αυτών των ε, προσαρτημάτων στη uh, um, you. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτά τα προσαρτήματα είναι ένα από τα προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη. Το πρόβλημα είναι ότι προκειμένου να αναλύσουμε το τι συμβαίνει στην πράξη, πρέπει κανείς να κάνει τη σωστή διάκριση μεταξύ των διαφορών προβλημάτων που προκύπτουν. Φαίνεται κάπως μπερδεμένο, αλλά θα προσπαθήσω να τα αποσαφηνίσω. Από τις συνομιλίες που είχαμε, μοιάζει κάποιες φορές η δικαιοπάροχη, δεν λέω ότι είναι ο κανόνας και ότι συμβαίνει σε κάθε μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά για να έχουμε μία γενική εικόνα στο μυαλό μας. Κάποιες φορές μιλάμε για αθέμητες ε, συμβασικές, συμβασικές σχέσεις. Κάποιες φορές είναι άδικοι οι δικαιοπάροχοι. Κάποιες φορές είναι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, όπως είπα. Α, όταν μιλάμε για προσαρτήματα, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, θα μπορούσε να είναι απλώς η άσκηση της συμβασιακής ελευθερίας, αλλά μπορεί να είναι όρος της σύμβασης που επιβάλλεται στον δικαιοδόχο αναλόγως με την πρακτική που αναπτύσσεται μεταξύ και τη σχέση μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου μπορεί να την εμπορική πρακτική. Είναι λίγο άδικο να το λέμε και χωρίς να το λαμβάνουμε υπόψη ε, ε, ότι εδώ υπάρχουν οι ρήτρες εμπιστευτικότητας και είναι κάπως κατανοητό. Και η τελευταία, η κυρία πίσω. Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι ένα προσάρτημα μπορεί να είναι κάποιε φορέ και προ όφελο ενό δικαιοδόχου, εξαρτάται από τι είδου ε, τέτοιο προσάρτημα είναι. Άκουσα όσα υπόθηκαν σήμερα το απόγευμα. Λέγομαι Ρωμάνα Έγκεμαν. Είμαι μάνατζερ από την Ολλανδική Ομοσπονδία των ε, Δικαιοδόχων και βλέπω πόσα υπόθηκαν σήμερα για τόσα καλό, τόσο καλά επιχειρηματικά μοντέλα. Δίνονται πολλές ευκαιρίες και στους δικαιοδόχους και στους δικαιοπαρόχους. Αλλά έχω ένα να πω. Σήμερα το απόγευμα είδαμε πόσο δυνατό είναι το λόμπι των δικαιοδόχων, ιδίως μάλλον των Ολλανδών και του τομέα της λιανικής τροφίμων. είναι ένα από τα βασικά θέματα του σημερινού απογεύματος. Εάν μιλούσαμε για συνεργασία και ισορροπία στι σχέσει δικαιοπαράγων δικαιοδόχων, ε, θα ήταν ε, πολύ θετικό αυτό. Αλλά μην βλέπουμε μόνο τι λένε οι Ολλανδοί και σκεφτούμε ότι είναι κάτι το πανευρωπαϊκό. Να μιλάμε για τη δικαιοδοσία. Καλό είναι, καλό να μιλάμε για την αυτορύθμιση και για τους κώδικες και πώς αναπτύσσονται, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με το σεβασμό των δύο πλευρών. Και υπόθεται κάτι άλλο πολύ σημαντικό για έναν κώδικα δεντολογίας που θα έπρεπε και αυτός ε, να γίνεται σεβαστός. Καλό θα ήταν εφόσον υπάρχει ο Ολλανδικός κώδικας. που έχει συνταχθεί από μια μικρή ομάδα και τώρα έχει ανοίξει και επηρεάζει όλες τις πλευρές, νομίζω σημαντικό είναι να υπάρξει συμφωνία όλων των εμπλεκομένων πλευρών, όχι μόνο των ε, ε, δικαιοπαρόχων. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται χρόνο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ε, πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά ομαδικά και με σεβασμό μεταξύ μας και πρέπει να γίνονται αυτά χωρίς να υπερισχύει μόνο ένα λόμπι. Ευχαριστούμε. Δεν σύμφωνα με τα επικριτικά σας σχόλια. Δώσαμε διπλό χρόνο ομιλίας στους ε, δίκαιο παρόχου για να μας εξηγήσει και τη δική τους θέση και το δικό τους κλάδο πιο αναλυτικά. Θέλω σύντομα να αντιδράσω, Ζανίν. Αν θες μάλλον Ζανίν να αντιδράσει, αυτά που υπόθηκαν για τον αδικό κώδικα. Άκουσα τις ε, παρατηρήσεις επανειλημμένως ότι μια ομάδα εργάστηκε κρυφίως και σιωπή. Δεν συμφωνώ, διότι συμμετείχαν εκπρόσωποι και των δικαιοπαρόχων και των δικαιοδόχων. Η κυρία Ένγεμαν, άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά τα των δικαιοπαρόχων σε αυτή την περίπτωση. Δημιουργήθηκαν think tank και στις, think tank και στις δύο πλευρές, στα δύο άκρα της Επιτροπής. Ξέρω πόσο καλά λειτουργήσε το κομμάτι των δικαιοπαρόχων και υπήρξαν συμβολές από πολλούς. Σκεφτήκαμε και το απόρριτο για την εμπιστευτικότητα, όπως εξήγησα προηγουμένως, με ε, το να αποφύγουμε την δημοσίευση στοιχείων στις εφημερίδες, ενώ ακόμα ε, σαν με τον κώδικα. Και ε, υπήρξε πολύ συμβουλευτική δραστηριότητα και από τι δύο πλευρές. Τώρα, τι έγινε καλύτερα στη μια πλευρά ή στην άλλη, με συγχωρείτε, δεν το έκανα εγώ. Ευχαριστώ. Είμαι βεβαίω ότι η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Επιτροπή έδειξε ιδιαίτερη υπομονή. Σα ευχαριστώ που μείνατε εδώ όλο το απόγευμα. Με μεγάλη χαρά θα σα δώσω το λόγο για να αντιδράσετε. Και έχω και μια ερώτηση. στι προηγούμενε αποφάσει του Κοινοβουλίου, σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, ζητούσαμε και από την Επιτροπή περισσότερη έρευνα εξέταση των ε, τρεχουσών πρακτικών. Έχει γίνει δουλειά στην Επιτροπή που θα μπορούσατε να μας την παρουσιάσετε, να μας πείτε τι να περιμένουμε και πώς πιστεύετε ότι η έκθεσή μου θα μπορούσε να είναι και για σας χρήσιμη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Θα αφήσω την δεύτερη ερώτηση να την απαντήσω ο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Growth αλλά θέλω να κάνω κάποια σχόλια για τα όσα ακούστηκαν σήμερα το απόγευμα και για τη μελέτη που μελέ, μελέτησε λεπτομερώς. Με ξέπληξε όντως ε, η μελέτη που, ε, μάλλον τα σχόλια που ε, λένε ότι δεν υπήρχαν, συμπερα... δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν μπορούσαν να βρουν τις συμβάσεις, αλλά παρόλα αυτά είχαν πάρα πολύ λεπτομερή συμπεράσματα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται να ισχύουν και τα δύο. Το πιο σημαντικό όμω είναι ότι η έκθεση βασίζεται σε μια βασική παρανόηση για, τον, ε, για τους κανόνες που υπάρχουν στην νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ο, η νομοθεσία ανταγωνισμού έχει να κάνει με την, ε, με την άδικη μεταχείριση στα, στις συμβατικές ε, σχέσεις. Το θέμα δεν είναι να ε, δούμε αν ε, κάποια, κάποια διάταξη ε, είναι πολύ αυστηρή για τον δικαιοπάροχο ή πολύ αυστηρή για τον δικαιοδόχο. Άλλο πράγμα μελετά η νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Επίσης ακούστηκε ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα της νομοθεσίας που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λέει η, μελέτη ότι από τη μία έχουμε την, τη δικαιοδοσία ε, του ανταγωνισμού και από την άλλη έχουμε την, ε, την νομοθεσία για, την, ε, για τις αθέμητες πρακτικές ή για, την, για το νυχικό δίκαιο. Αν δεν, η νομοθεσία αν δεν ήταν έτσι όπως είναι, δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την νομοθεσία περί ανταγωνισμού και στο τέλο και οι δικαιοπαροχοί και οι δικαιοδόχοι, αλλά ούτε και οι καταναλωτέ δεν θα μπορούσαν να έχουν οποιοδήποτε όφελο. Το να λέτε στου πελάτε σα ή στα μέλη των ομοσπονδιών σα ότι θα πρέπει να πάνε στο δικαστήριο και να, για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ε, στα πλαίσια τη νομοθεσία του ανταγωνισμού, ουσιαστικά δημιουργείται κόστος για τους νομικούς χωρίς να υπάρχει ε, περίπτωση να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα γιατί τα κριτήριά σα ήταν πολύ υψηλά ή ήταν πολύ ε, ε, απαιτητικά. Πάτε στο δικαστήριο και λέτε ναι, αλλά δικαστήριο πρέπει να μου λύσετε αυτό το πρόβλημα. Όχι, ε, όχι ως την πρακτική, ως, αλλά ως θέμα ανταγωνισμού. Ο, ο δικαστής θα σα ρωτήσει πώς περιορίζεται ο ανταγωνισμός εδώ, πού είναι το πρόβλημα, πώ δεν μπορεί ο δικαιοδόχο να μπει στην αγορά γιατί περιορίζεται ο ανταγωνισμό επειδή οι απαιτήσει για τι επιδόσει σα ήταν πολύ υψηλέ. Οπότε θα πληρώσετε πάρα πολλά τέλη στον νομικό και τελικά δεν θα λύσετε και το πρόβλημά σα. Και μετά το επόμενο ερώτημα είναι, θέλουμε, όπω είπαν μερικοί από εσά, να αλλάξουμε τους στόχους του στόχου τη νομοθεσία ανταγωνισμού. Να βάλουμε δηλαδή διαφορετικού στόχου, να να πρέπει να πετύχει άλλα πράγματα. Και αν το κάνουμε, γιατί να μην δούμε και την επίπτωση στον, στην απασχόληση και τι γίνεται με τις συμβατικές σχέσεις. Γιατί να μην δούμε τις ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών. Στο τέλος θα έχετε μία πολιτική αναποτελεσματική για τον ανταγωνισμό που θα είναι αναποτελεσματική κυρίως επιζήμια για τις μικρές επιχειρήσεις. Όταν αλλάξαμε το 99 τους κανόνες, ξέρετε ποιοι ήταν αντίθετοι με τους ε, νέους κανόνες. Οι, ε, οι και οι, οι Γιατί θα είχαν ε, πολύ περισσότερε δυνατότητε να έχουν εξαιρέσει χωρί να υπάρχουν κατόφλια όπω υπήρχαν στην παλαιά νομοθεσία. Αυτό νομίζω ότι είναι ο ρόλο τη ε, νομοθεσία. Το επόμενο ερώτημα είναι, θα πρέπει να υπάρχει άλλη νομοθεσία να παρέμβουμε εάν υπάρχουν ε, αθέμητες πρακτικές. Εδώ ειλικρινώς πρέπει να σας πω ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα δεδομένα από τα να αναφέρεστε μόνο στον φόβο που υπάρχει. Και μετά το ερώτημα είναι σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι κάνουμε. Και εδώ θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να... γιατί αυτός είναι εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης που είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς ε, για τις σχέσεις ε, μεταξύ επιχειρήσεων εργάζομαι. Εδώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και, του, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εμπορικές πρακτικές στην, ε, στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα και θα ήθελα να πω και εγώ τη δική μου άποψη για το πώς βλέπουμε το μέλλον της δικαιοχρησίας. Καταρχάς, το βασικό πρόβλημα νομίζω ότι είναι ε, συγκρίσιμο στις δύο αυτούς τομείς. Υπάρχουν πολλές ανισορροπίες, υπάρχουν αθέμητες πρακτικές και υπάρχει και ο φόβος που είναι κατανοητός. Αυτό που βλέπουμε στην αλυσίδα τροφοδοσία είναι κάποιε θελοντικέ πρωτοβουλίε που μπορούν να λειτουργήσουν. Βέβαια, είναι μακρά η διαδικασία και δύσκολο ο δρόμο, αλλά νομίζω ότι αυτά τα αυτορυθμιστικά προγράμματα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και στην δικαιοχρησία. Και το σημαντικό είναι ότι είναι διμερής η διαδικασία αυτή. Ο μονομερής λοιπόν κώδικας οντολογίας που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δικαιοχρησία μάλλον δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Νομίζω ότι οι διατάξει που έχουμε στις κατοχώρε, που είναι διμερής διαδικασία είναι πολύ, πολύ πιο πολλά υποσχόμενοι. Οπότε σα ευχόμαστε καλή επιτυχία με το Ολλανδικό μοντέλο, γιατί πραγματικά και εμεί περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν και, οι δύο, ε, και τα δύο μέρη να εμπλέκονται με ίσο και δίκαιο τρόπο. Και βεβαίως υπάρχει ανάγκη να οργανωθούν ε, οι δικαιοδόχοι αποτελεσματικά έτσι ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν ένα τέτοιο κώδικα όχι μόνο στο Ολλανδικό, στην Ολλανδία αλλά και σε, άλλες, ε, σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ιστορική αγορά. Υπήρξαν πολλά σχόλια σήμερα για το τι γίνεται με τα προβλήματα στην δικαιοχρησία και πώς αυτά εμποδίζουν την ιστορική αγορά. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί εγώ στη μελέτη δεν είδα πολλές αποδείξεις για τα προβλήματα που δήθεν προκαλούνται στην εσωτερική αγορά και ε, βλέπω ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι... Δεν, δεν είδα μάλλον στοιχεία που να δείχνουν ότι όντω και τα διασυνοριακά, οι διασυνοριακέ εμπορικέ σχέσει ε, επηρεάζονται. Οπότε καλό είναι να λέμε ότι να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε έτσι τόσο γενικόλογα. Αυτό που βλέπουμε όταν μπαίνουμε σε τέτοιε λεπτομέρειε είναι ότι όλε αυτέ οι πολυεθνικέ οργανώνονται με τέτοιο τρόπο που οι, ε, τοπικές, ε, οι τοπικοί δικαιοδόχοι του, στη μεγάλη του πλειοψηφία, ε, δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τι ε, αποδείξει που υπάρχουν. Και αυτά που ακούσαμε κυρίω είναι εσωτερικά προβλήματα. Οπότε στα πλαίσια και τη επικουρικότητα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ε, ε, καταλήγουμε σε συμπεράσματα γενικά που λένε ότι πρέπει τα προβλήματα να ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν υπάρχει κίνδυνο για την εσωτερική αγορά. Αλλά Τώρα βρισκόμαστε ε, στην ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσπαθεί να έχει πολύ πιο, καλύτερους, πιο, καλύ, πιο καλούς κανόνες διαχείρισης και στα πλαίσια αυτά προσπαθεί να είναι πολύ προσεκτική. Πρέπει λοιπόν να το δούμε. Όπως είπα η μελέτη, δεν την κρίνω για τα συμπεράσματά της αλλά δεν μας αποδείχνει ότι υπάρχει αντίκτυπος ε, διασυνοριακός ή ότι υπάρχουν ε, διαρθρωτικά προβλήματα για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μια ερώτηση που την ξανακάνουμε. Ήταν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου στο παρελθόν. Και τότε σας ζητούσαμε, εσείς η Κομισιόν να κάνετε μία μελέτη για τις επιχειρηματικές στρατικές ε, στον τομέα της δικαιοχρησίας. σχολιάσατε τη δική μας μελέτη, τη μελέτη που έγινε για εξονομώσεις του Κοινοβουλίου. Αλλά εσείς τι υλικό έχετε για να μας βοηθήσετε, ούτω ώστε να σχηματίσουμε ε, μία γνώμη και να φτιάξουμε μια εμπεριστατωμένη έκθεση. Καταρχάς είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ε, είχαμε τρία άτομα που ασχολούνται με αυτό το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και τα τελευταία δύο χρόνια ασχολιόμασταν κυρίως με την τροφική αλυσίδα. Τον Ιανουάριο του 2016 ετοιμάσαμε μια έκθεση, η οποία ήταν πολύ εμπεριστατωμένη και ανέλυε το κανονιστικό πλαίσιο και στα 28 κράτη-μέλη και κάναμε και μια ανάλυση ε, όλων των πρωτοβουλειών που υπάρχουν στην τροφική αλυσίδα. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώ θα ξοδέψουμε του ε, πόρου μα και του ανθρώπινου πόρους μα, γιατί υπάρχουν διάφοροι τομεί που ενδιαφέρουν, ας πούμε, διάφορους stakeholders ε, και όπου υπάρχουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές ο τομέα των αυτοκινήτων, α πούμε, έχει προβλήματα. Ε, πολλοί τομεί έχουν προβλήματα, κάπου θα πρέπει να εστιάσουμε τις προτεραιότητες και να αποφασίσουμε που θα δώσουμε, ας πούμε, βαρύτητα. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και άλλα δεδομένα. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Από τις επαφές που είχαμε με άλλους τομείς, μπορώ να σας πω ότι ε, μια και μία διαφάνεια έλεγε να μην έχουμε τομιακή προσέγγιση. Έχω να σας πω ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, τέτοια θέματα, όπως αυτά που αναφέρατε εσείς, υπάρχουν και σε άλλους τομείς. Αν δείτε, ας πούμε, αν μιλήσετε με ζηθοποιούς, θα δείτε ακριβώς τα ίδια προβλήματα με αυτά που έχετε εδώ. Τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες συζητήσεις. Σε ποιο βαθμό, ας πούμε, η ζηθοποιοί υποτίθεται ε, ότι μπορούν ε, να δεσμεύουν ή να μην δεσμεύουν, ας πούμε, τους ιδιοκτήτες των pub, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Αν νομίζετε ότι αυτά αφορούν δικά τη δικαιοχρησία, πλανάστε. Εάν η δικαιοχρησία είναι θέμα ανταγωνισμού, και, το, και προσπάθησε η μελέτη να εξετάσει τις υποθέσεις που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν ελάχιστες και όταν υπήρχαν αφορούσαν τις ε, κάθετες, ε, τους κάθετους περιορισμούς, κάποιους περιορισμούς που έθεταν οι δικαιοπάροχοι στους δικαιοδόχους και κάποια όρια που τους έθεταν στις τιμές, ότι θα φτάσεις μέχρι εκεί δεν μπορείς να πέσεις πιο κάτω ας πούμε. Και επίσης ε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ειδικού κανόνες που θα εξαιρούν τη δικαιοδοσία από τους κανόνες ανταγωνισμού. Δεν θέλω να φτάσω συμπεράσματα για την έκθεση ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε βαθμιδών. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι από τη μία δεν πρέπει να έχουμε τίποτα συγκεκριμένο ε, για τη δικαιοχρησία στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού. Και από την άλλη, μα λέτε εσεί να μην κάνουμε τίποτα. Έτσι. Γιατί μια χαρά είναι η κατάσταση. Τότε, εντάξει, δεν με βοηθάτε και πολύ. Καλύτερα να μου λέγατε, εντάξει, θα δούμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα, το, θα, θα κάνουμε ένα follow-up, θα κάνουμε κάποιε έρευνε, θα, κάποιο, θα εξετάσουμε την κατάσταση, θα δώσουμε μια συνέχεια τέλο πάντων. Και μπορούμε να σα βοηθήσουμε, αφού ας πούμε συγκεντρώσετε αυτέ τι πληροφορίε, να σα βοηθήσουμε αυτέ τι πληροφορίε. Αλλά η απάντησή σα, μην κάνετε τίποτα, μην κάνετε τίποτα για την δικαιοχρησία, δεν νομίζω ότι μα αρέσει. Δεν είναι η σωστή απάντηση που θα, πρέπει να μας δώσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ο συνάδελφος, αν κατάλαβα καλά τι είπε, είπε ότι δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα αθέμητων πρακτικών στη δικαιοχρησία, αλλά ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πει θέλω να ρυθμίσει ε, θέλουν να ρυθμίσω ένα τομέα, θα μα πούνε αμέσω γιατί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιο είναι το διασυνοριακό στοιχείο, η διασυνοριακή διάσταση. Γιατί χρειαζόμαστε έναν ενωσιακό κανονισμό και να τα αφήνουμε όλα τα κράτη-μέλη. Επομένω, χρειαζόμαστε αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εσωτερική αγορά, ένα διασυνοριακό πρόβλημα. Πριν ζητάτε από την Κομισιόν να ρυθμίζει κάποια πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αμέσω, αλλιώ αμέσω αντιδρούν οι πολιτικοί. Και όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά βεβαίω και στην Ολλανδία, θα μα πούνε, ότι γιατί δεν ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το θέμα. Πρόεδρο, γι' αυτό ζητάμε ω Κοινοβούλιο από την Κομισιόν να διερευνήσει τον τομέα αυτό. Και δεν το έκανε. Και μα είπε δεν το έκανε λόγω έλλειψη πόρων. Όπω και εγώ. Προσπαθώ να μην προδικάσω τίποτα, έτσι, να μην φτάσω σε συμπεράσματα πρόωρα, Νομίζω ότι είναι πολύ ομό για την Κομισιόν και πολύ απότομο, έτσι, χωρίς ε, στοιχεία, να έχει και άποψη για το τι είναι σωστό και τι όχι. Κάναμε την ίδια συζήτηση για το λιανεμπόριο στον τομέα των τροφίμων. Τέλος πάντων, το είπα και από ότι δεν πρόκειται τώρα να πω τίποτα άλλο. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μας. Αλλά να σας πω κάτι σε όλους να αφού σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας. Ως μελλοντικός συγητής θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτα αμερόληπτος, να λάβω υπόψη όλες τις συνεισφορές όλων των πλευρών προς το παρόν. Δεν έχω σχηματίσει άποψη. Αντίθετα από την Κομισιόν, η οποία μας λέει αυτό πρέπει να γίνει και όχι το άλλο, εγώ θέλω να τα δω όλα. Ανοιχτά τα μάτια έχω, ανοιχτό το μυαλό θα μιλήσω με όλους, τους εκπροσώπους των δικαιοπαρόχων, των δικαιοδόχων, τις ενώσεις τους, ε, τους δικούς μας ερευνητές. Θα ξαναδιαβουλευτώ με όλους και σε διμερή βάση. Και στην έκθεση που ούτως ή βραχία πρέπει να είναι, εξάλλου οι εκθέσεις ιδίες πρωτοβουλίες είναι πάντα πολύ σύντομες, στην έκθεση λοιπόν θα, προσπαθήσω να φτάσω στα συμπεράσματα. Έχουμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Ελπίζω να σας ξαναδώ κάποιους από εσά και να καταλήξω σε κάτι το οποίο θα κινείται προς την κατεύθυνση και προς αυτό το πνεύμα που μας περιέγραψε η Ομοσπονδία EFF τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, να λάβουμε υπόψη μα τη σημασία τη δικαιοχρησία και στην εσωτερική αγορά, το ότι μπορεί να υποφελήσει η δικαιοχρησία για την εσωτερική αγορά και μέσα σε αυτό το έτσι γενικό πλαίσιο θα κινηθώ. Αυτά. Ευχαριστώ για όλες τις α, συνεισφορές σας. Ήταν μια συζήτηση, η εναρκτήρια θα έλεγα, συζήτηση μιας μακράς διαδικασίας. Γεια σας.